Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς θερμότατα στην ακρόαση του υποψηφίου επιτρόπου για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών. Καλωσορίζω θερμότατα τον κύριο Τζον Ντάλι. Καλώς ορίσατε στην επιτροπή μας. Η ακρόαση αυτή διεξάγεται από κοινού με την Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς και την Επιτροπή Γεωργίας και καλωσορίζω τους συναδέλφους από τις δύο αυτές επιτροπές, ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Επιτροπής εσωτερική Αγοράς, τον κύριο Μάλκολμ Χάρμπορ. Καλωσορίσατε θερμά για την κοινή μας ακρόαση. Στι επόμενε τρει ώρε θέλει να αποκομίσει η Επιτροπή και οι βουλευτές άποψη για τις ικανότητες και τα προσόντα γενικά του υποψηφίου για ένα τέτοιο ε, πόστο, αν έχει ευρωπαϊκές πεπιθήσεις και ανεξαρτησία προσωπική από οποιαδήποτε συμφέροντα για να ασκήσει τα καθήκοντά του και το Κοινοβούλιο επίσης αξιολογεί τις ειδικέ γνώσεις του υποψηφίου ως προς το χαρτοφυλάκιο και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Κάτι που είναι σημαντικό γενικά στην πολιτική και ιδιαίτερα ακόμα στην ευρωπαϊκή πολιτική για να απευθύνεται κανείς και να φτάνει μέχρι τους πολίτες και την κοινή γνώμη. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν που έχουμε για να, πριν ψηφίσει το Κοινοβούλιο για τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε λάβει το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία διαξαγωγής. Θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουμε ένα λεπτό για τις ερωτήσεις, δύο λεπτά για τις απαντήσεις, 45 δευτερόλεπτα για συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό και πάλι για συμπληρωματική απάντηση. Έτσι έχουν οι κανόνες του παιχνιδιού και παρακαλώ να τηρούν όλοι τους χρόνους σας. Επίσης, Όποιο είναι απόνοτο του δίνουμε το λόγο, χάνει τη σειρά του και ελπίζω να συμμετέχετε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολόκληρης. Κύριε Τάλη, τα τελευταία 20 χρόνια ε, είχατε διάφορα καθήκοντα και ε, αξιώματα στην κυβέρνησή σας, ε, οικονομικά, οικονομία, εξωτερική πολιτική, κοινωνική πολιτική και τώρα καλείστε να εκπροσωπήσετε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 500 εκατομμύρια πολίτες, ε, ε, να ε, υπομειστείτε το χαρτοφυλάκιο της υγείας, προστασίας της δημότητας υγείας και του καταναλωτού. Αυτοί είναι δύο τομείς που θεωρούν πάρα πολύ σημαντικούς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο το Κοινοβούλιο, αλλά και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αξιολογούν ως μεγάλη προτεραιότητα. Ε, διάβασα τις γραπτές σας απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά γενικές. Και ελπίζουμε τώρα στις επόμενες τρεις ώρες να δώσετε ένα προσωπικό τόνο και το όραμά σας, το πολιτικό όραμα, να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πώς θα προσανατολιστείτε για την επόμενη θητεία, την επόμενη πενταετία. Και περνούμε αμέσω στην ουσία του θέματος. Έχετε το λόγο για την εισαγωγική σας παρουσίαση. 10 λεπτά παρακαλώ. Good morning, ladies and Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να συμμετάσχω σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Ένα θεσμικό όργανο το οποίο μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας αναλαμβάνει μεγαλύτερες ευθύνες για την προώθηση των αξιών και του ευρωπαϊκού οράματος. Ήμουν μέλος της Βουλής της χώρας μου για πάνω από δύο δεκαετίες. Στα τρία τέταρτα του χρόνου αυτού ήμουν και μέλος της κυβέρνησης. Αυτό μου δείχνει μια βαθιά κατανόηση της διάδρασης ανάμεσα σε Βουλή και στην εκτελεκτική εξουσία και τον σεβασμό των απόψεων του Κοινοβουλίου. Έχω υπηρετήσει και ως μέλος της κυβέρνησης της χώρας μου για πολλά χρόνια κυρίως στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, προωθώντας μεταρρυθμίσεις και σεβόμενος το κοινοτικό και εκτιμένο. Όμως, τη μεγαλύτερη ευθύνη ένιωσα τα τελευταία 18 μήνες που ήμουν υπεύθυνος για θέματα υγείας. Αυτό με έφερε πιο κοντά στους ανθρώπους και στην πρώτη γραμμή για να δώσω την καλύτερη υπηρεσία στους πολίτες και να καλύψουμε τα χάσματα των γενεών και των φίλων. Αυτό μου έδωσε την ικανοποίηση να, ικανοποιήσω τις φιλοδοξίες μου ως πολιτικού άντρα. Τις επόμενες τρεις ώρες θα θίξουμε πολλά θέματα. Θα ανταλλάξουμε πολλές απόψεις. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά μπορούν να εγγραφούν σε ένα μόνο θέμα. Τον κόσμο. Τώρα επιτρέψτε μου να θίξω ορισμένα θέματα στη μητρική μου γλώσσα. Il paziente Πρώτα απ' όλα οι ασθενείς, πρώτα απ' όλα οι καταναλωτές. Αυτό θα είναι η κατευθυντήρια γραμμή της εργασίας μου, εάν μου δώσετε την ευκαιρία να αναλάβω τα καθήκοντα του Επιτρόπου. Θα είμαι ανεξάρτητος, αντικειμενικός στην αξιολόγηση των διαφόρων θεμάτων που, για τα οποία θα είμαι υπεύθυνος. θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία που έχω για δημιουργία συμφωνιών και την εμπειρία μου από τους διάφορους τομείς για να προσθέσω αξία στα διάφορα προγράμματα που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν αλλά και στα προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν σύντομα. Το όραμά μου είναι το όραμα ενός Ευρωπαίου πολίτη που θα έχει μια μακρύτερη και υγιέστερη ζωή ακριβώς γιατί έχουν υγιέστερη διαβίωση, θα έχουν πρόσβαση σε πιο υγιή είδη διατροφής και θα έχουν υψηλής ποιότητας περίθαλψη και φάρμακα. Έχω το όραμα ενός σωστά ενημερωμένου καταναλωτή που μπορεί να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για τα προϊόντα που καταναλώνει. Ένας καταναλωτής ο οποίος θα κατευθύνει όχι μόνο τη ζωή του, αλλά θα μπορεί επίσης και να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων. Οι καταναλωτές μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές σε τομές όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, την ευημερία των ζώων, την υγεία. Είμαι δεσμευμένος για να εξασφαλίσω ότι οι καταναλωτές μας θα εξακολουθούν να έχουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ειδών διατροφής. Και θεωρώ ότι όλοι αυτοί προσπαθούμε να επιτύχουμε και να θέσουμε τα πρότυπα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Η καινοτομία επίσης είναι σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου μας και έχουμε μεγάλη δυνατότητα να καινοτομήσουμε και στις ζωοτροφές, στις ε, ιατρικό εξοπλισμό, φαρμακευτικά προϊόντα και το καθεξής. Μιλάμε εδώ για την δυνατότητα καινοτομίας προς όφελος των καταναλωτών μας και των πολιτών μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, για τη δημόσια υγεία, τώρα που έχουμε μείωση των προϋπολογισμών, τίθεται το θέμα της βιωσιμότητας των συστήματων υγείας. Για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα θα πρέπει να εστιμάσουμε την προσοχή μας στην πρόληψη. Πάνω το 97% ε, των δαπανών στην Ευρώπη πάνε για την περίθαλψη και το 3% μόνο για την πρόληψη. Θα ήθελα να αντιστρέψω αυτή την ανισορροπία. Η πρόληψη είναι επένδυση και έχει μεγάλα αποτελέσματα στο μέλλον. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να επιτύχουμε βιωσιμότητα στην υγεία και να έχουμε έρευνα σε ό,τι αφορά τις καρδιοαγγειακές ε, ασθένειες, τον καρκίνο και τις άλλες ασθένειες και να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα, την κατάχρηση νοπνευματοδών, την παχυσαρκία που φάνηκε ότι είναι μεγάλες αιτίε για την νοσοκομιακή περίθαλψη εκατομμυρίων ασθενών κάθε χρόνο. Βασικό τμήμα της του οράματος είναι η πρόσβαση των πολιτών, σε ό, όλων των πολιτών, σε έγκαιρη ε, περίθαλψη, καλή περίθαλψη και ε, ικανοποιητική τιμή για τα φάρμακα. Δεν υπάρχει λόγος οι φτωχοί να έχουν κακή υγεία. Γι' αυτό θα συνεργαστούμε με την Ισπανική Προεδρία, με το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο για να βρούμε μια λύση για την περίπτωση των ασθενών στην διαβεθυσινοριακή περίθαλψη. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης και την ε, που ε, προσφέρονται από τη συμπερίληψη αυτών των θεμάτων στο χαρτοφυλάκιό μου. Μπορούμε να έχουμε έτσι καινοτόμες λύσεις για την έρευνα και να βρέσουμε νέες ε, περιθάλψεις για τους ασθενείς στην Ευρώπη. Θέλουμε να καλύψουμε τα χάσματα της ε, ανισορροπίας για την υγεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει 14 έτη διαφορά στο προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη από τη μία περιοχή στην άλλη και αυτό είναι εις βάρος της συνέπειας και της συνοχής της Ευρώπης και είναι απώλεια του οικονομικού μας δυναμικού. Αυτό θα πρέπει να είναι σημαντικός στόχος που θα πρέπει να θέσουμε αυτούς για να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Η ενημέρωση των ασθενών είναι άλλο ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται. Πιστεύουμε ότι ο ασθενής θα πρέπει να έχει πρόσβαση για συντακολογούμενα φάρμακα που είναι στην αγορά η συμπερίληψη του φάρμα στο χαρτοφυλάκιό μου μας δίνει και δυνατότητα να εκτάσουμε την πρόταση ξανά. Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια συμπεριλαμβάνει και τις δράσεις κατά παρεποιημένων φαρμάκων που προλα... στο ίντερνετ. Προτείνω να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στα θέματα της παραποίησης φαρμάκων και φαρμακοεπαγρύπνησης για την πολιτική των καταναλωτών θα διατηρήσω την μεγάλη σημασία που έχουν τα θέματα των καταναλωτών όπως έγινε τα τελευταία χρόνια. Τα θέματα καταναλωτών αφορούν πολλά αχαρτοφυλάκια και εγώ έχω ως βασικό ρόλο να προωθήσω τη διάσταση των καταναλωτών σε όλα αυτά τα θέματα και συζητήσεις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ενιαία αγορά σωστά υπηρετεί τον καταναλωτή μέσω καλής πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά σε, με καλή διαθεσιμότητα και τιμές. Πρέπει να δούμε το πώς η αγορά υπηρετεί τους καταναλωτές και ποιες δομές πρέπει να αλλάξουν για να γίνουν αυτά καλύτερα. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενισχυμένο scoreboard για τους καταναλωτέ. Σκοπεύω να κάνω συνεχείς έρευνες για να ενισχύσω τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε εξουσία στον καταναλωτή δίνοντάς του επιστημονικά βασιζόμενη γνώση. Ταυτόχρονα οι καταναλωτές πρέπει να έχουν γρήγορη και αποτελεσματική ε, διόρθωση και γι' αυτό θα έχουμε συνολική πρόταση και επανεξέταση όλων των προτάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την ασφάλεια των ειδών διατροφής. Θέλω να εξασφαλίσω ότι η νομοθεσία μας θα έχει την ισορροπία παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή με ε, αποτελεσματικά οικονομικό τρόπο. Είναι ο τομέας των ειδών διατροφής ο μεγαλύτερος εργοδότης και είναι ο κρίκος ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή. Κανένας δεν έχει να κερδίσει τίποτα από χαμηλά επίπεδα ασφάλειας στα είδη διατροφής. Χρειαζόμαστε αυτά τα επίπεδα υψηλής ασφάλειας να είναι θετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στη διεθνή αγορά. Τα πρότιμά μας είναι προ, προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτό με τη σειρά του είναι στην υπηρεσία των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών και της βιομηχανίας μας. Μας δείχνει η εμπειρία ότι θέτοντας πρότυπα οδηγούμε τη βιομηχανία μας να καινοτομήσει περισσότερα και ταυτόχρονα δημιουργεί μεγαλύτερης ε, προστιθέμενης αξίας προϊόντα Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο να εξασφαλίσουμε επίσης ότι όλα τα ζώα θα υποφεληθούν από την σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων. Επιπλέον έχω την πρόθεση να σας υποβάλω μία έκθεση για την μεταφορά των ζώων σε ένα χρόνο και τις πολιτικές που θα αναλάβουμε στον τομέα αυτό. Λάβαμε το μήνυμά σας, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Thank you very much. First... σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά ακούω ε, τόσο μεγάλο μέρος λόγου στα Μαλτέζικα. Ε, σας έδωσα και ένα λεπτό περισσότερο γιατί έγινε και η μετάφραση ταυτόχρονα. Ευχαριστώ για την εισαγωγική σας ομιλία. Θα αρχίσουμε τον πρώτο γύρο με τους ε, συντονιστές και πρώτος ο, Πέτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφιοι Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την εισαγωγική σας ομιλία που έδειξε ότι έχετε εμπειρία αλλά και έχετε και πεπραγμένα στον τομέα της υγείας. Εγώ θα ερωτήσω σχετικά με τον ρόλο του ασθενούς στην ε, πολιτική υγείας της Ευρώπης. Είπατε στις γραπτές σας απαντήσεις ότι θέλετε να υποστηρίξετε και τους ανεξάρτητους ασθενείς από το Health Action Program, το οποίο έχει καλή χρηματοδότηση. Έχετε και άλλες ιδέες σχετικά. Δεύτερο, η ενημέρωση για τους ε, ασθενείς σχετικά με τα φάρμακα διεξάγονται εντατικές συζητήσεις τώρα σχετικά με την πρόταση του Επιτρόπου Φερχόγγεν. Υπάρχει όμως και η συνένεση ότι η παρούσα κατάσταση με την ελληπή ενημέρωση δεν είναι ικανοποιητική και χρειάζεται περισσότερη ανεξάρτητη ενημέρωση. Μπορείτε να φανταστείτε σε συνδυασμό της προσπάθειάς σας με, με τις δικές μας προσπάθειες να ενισχυθούν οι ανεξάρτητες πληροφορίες, η ανεξάρτητη ενημέρωση των ασθενών να ενισχυθεί λοιπόν η προσπάθεια αυτή μέσα από μια προσπάθεια δική σας και δική μας. Απάντηση. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες ασθενών, πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι οι ομάδες αυτές ασθενών έχουν σημασία για την ανάδραση, για το feedback και για μια συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης και είναι απαραίτητο να διατυπωθούν εδώ ιδέες. Είναι σημαντικό στην διαδικασία λήψης αποφάσεων να δούμε τα πράγματα και μέσα από την οπτική του ασθενούς για τις πολιτικές αυτές. Και αυτό επομένως θα αποτελέσει δική μας υποχρέωση να διασφαλίσουμε ώστε οι ομάδες αυτές ασθενών να υποστηριχθούν επαρκώς. Συμφωνώ μαζί σας. Πάλι βεβαίως θα, έχουμε, θα έχω να διαχειριστώ προϋπολογισμό που δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλος της υγείας. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και πιέσεις για τη χρηματοδότηση από τον προπολογισμό τέτοιων ομάδων και σίγουρα θα χρειαστεί να αναζητήσουμε νέε ιδέε για να δούμε πώ μπορεί να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτή. Θα είμαι ανοιχτό στι ιδέε ε, τι δικέ σα και ίσω μπορώ να συμβάλλω με τη δική μου εμπειρία στην διαμόρφωση τέτοιων προγραμμάτων, τέτοιων μηχανισμών για την υποστήριξη των ε, ομάδων αυτών ασθενών και καταναλωτών εν τέλει. Υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίσουμε, και αυτό είναι σημαντικό, την ανεξαρτησία τους. Εν τέλει, και αυτός ίσως είναι ένας τρόπος, εάν δηλαδή μπορέσουμε να ιδρύσουμε κάποια συστήματα, ώστε οι πόροι που καταλήγουν στις ομάδες αυτές ασθενών να μην έρχονται απευθείας από τη βιομηχανία, αλλά μέσα από κάποια συστήματα που μπορούμε να φτιάξουμε μαζί, εσείς και εμείς, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να ε, το φτιάξουμε σε συνεργασία. Γιατί αυτό θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε, σας ευχαριστώ για την ακριβή απάντηση. Τα δύο λεπτά που έχω ακόμη δεν μου επιτρέπουν να έλθω στην ενημέρωση των ασθενών, γι' αυτό έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Ποιες αλλαγές και ιδίως συμπληρώσεις της προτάσεως του κ. Φερχόγγεν θεωρείτε ότι μπορείτε να κάνετε. Δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας βέβαια διαμιάς, αλλά έχουμε τώρα αυτό το πακέτο, την δέσμη μέτρων φαρμακολογίας, με τρεις βασικούς πυλώνες για την ε, ε, ενημέρωση των ασθενών και άλλα. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι πυλώνες είναι σημαντικοί. Δύο από αυτά δεν είναι αμφιλεγόμενα. Η πρότασή μου είναι να προχωρήσουμε με τα δύο αυτά στοιχεία, αν θέλετε, όσο γίνεται συντομότερα, έστω και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε το θέμα της ενημέρωσης του ασθενούς. Τώρα που τα φάρμακα έχουν μπει μέσα στο χαρτοφυλάκιο της υγείας, σας διαβεβαιώ ότι θα επαναξιολογήσουμε την δέσμη αυτή του κ. Βερχόγγεν και θα βάλουμε μέσα περισσότερο την οπτική γωνία του ασθενούς στις προτάσεις και μετά θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες συζητήσεις μαζί σας. Γνωρίζω ότι και εσείς συζητείτε την δέσμη αυτή στο Κοινοβούλιο και ε, θα τίνω βέβαια νους στα όσα έχετε να μου πείτε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Μακάβαν. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Μιλήσατε για τους ανθρώπους και για τη σημασία του Ευρωπαίου πολίτου. Εδώ εμείς συζητούμε και μας παρακολουθούν τώρα στο διαδίκτυο. Και η σοσιαλιστική ομάδα ακούει ερωτήσεις του κοινού που αναφέρονται στο κάπνισμα, αναφέρονται στο ενόπνευμα, στην μεταφορά των ε, ζώων, στις μεταφορές των ζώων δηλαδή, στην παχυσαρκία. Ποιες προτεραιότητες θα επιλέξετε, ποια θα θέλατε να είναι η κληρονομιά σας μετά από μια πενταετία ως ε, επίτροπος. Περισσότερο να ρίξετε το βάρος σας, για παράδειγμα, στην ευημερία των ζώων σε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να είμαι ο Επίτροπος που θα δείξει σκληρή στάση σε όλα τα θέματα αυτά. Γιατί είναι τα θέματα που όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία είναι πράγματα τα οποία προκαλούν δεινά. Αν αναγκάζουν του ανθρώπους να καταφεύγουν στα νοσοκομεία για εκατομμύρια, μιλώ για εκατομμύρια πολίτε. Εγώ θα ήθελα πάντω να με θυμούνται για το ότι έφερα τη συζήτηση αυτή στα σχολεία. Θεωρώ ότι Εν τέλει αυτό είναι ζήτημα δεξιοτήτων της ζωής. Δηλαδή του να μπει η παιδεία στις επιλογές ζωής που κάνει ο καθένας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του νέου για το τι είναι τελικά καλό για τον καθένα. Και μετά θα δούμε και τα άλλα, ε, επισημάνσεις, ετικέτες κτλ. Αλλά εκεί μπαίνουν αυτά, εντάσσονται σε αυτό τον βασικό πυλώνα. Και όσο νωρίτερα αρχίσουμε εκπαιδεύοντα τα παιδιά μας, τόσο καλύτερα. Θα αρχίσουμε να μιλούμε για την ζημιά που κάνει ο καπνός, για παράδειγμα, για τη ζημιά που κάνει η κατάχρηση νοπνεύματος, για το τι πρέπει να τρώει κανείς και πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του κάνοντας σωστές επιλογές σε ό,τι καταναλώνει για παράδειγμα σε λίπη, σάκχαρα κτλ. επίση η καλή άσκηση. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητα. Κύριε Μακάβαν, αρκεί η ενημέρωση. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε, έχουμε ενημέρωση για τους κινδύνους του αλκοόλ, για τους κινδύνους του καπνίσματος. Ορισμένοι λένε, μα είναι το κράτος γκουβερνάντα. Τι δράσεις θα αναλάβετε για να πείσετε και αυτούς. Η ενημέρωση των πολιτών δεν είναι μόνο θέμα του κράτους. Το κράτος είναι ε, διαπαιδαγωγή. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε νομοθεσία κατά ή σε κάθε λεπτομέρεια αλλά να προωθήσει την ενημέρωση και να σταχυολογήσει τις βέλτιστες πρακτικές από τις διάφορες χώρες μέλη και να προσπαθήσει να τις ε, εντάξει όλες αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και σε αυτά στις πολιτικές που θα ασκήσει εν τέλει. Εκεί θα χρειαστεί ανάληψη δράση και εκεί βεβαίω χρειάζεται και χρηματοδότηση. Χρειάζονται χρήματα. Επανέρχομαι βέβαια στο ίδιο θέμα. Αν θέλουμε να πετύχουν τα πράγματα αυτά, πρέπει όχι απλώ να συνεχίσουμε να, παρα... να παραπονούμαστε για το ότι δεν γίνεται τίποτα, αλλά να βρούμε πραγματικά πόρου δημοσιονομικού για να μπορέσουμε να τα πληρώσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Το κόστο των συστημάτων υγεία είναι υψηλό και αυξάνεται ένα μικρό ποσοστό από όλη αυτή τη χρηματοδότηση να πάει για την πρόληψη, την ενημέρωση. Νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει πολύ. Η κυρία Μπλεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, προηγουμένως είπατε ότι δίδεται μεγάλη σημασία στην πρόληψη και χαίρομαι γι' αυτό, διότι στις προτεραιότητες σας δεν το είχα αντιληφθεί ως προτεραιότητα η, ψυχική, η, υγεία, η και η δημόσια υγεία είναι πολύ σημαντική και επίσης και η διατροφή. Ε, εδώ έχετε κληρονομήσει ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα που είναι οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί και θα πρέπει να βασίζεται ε, πάντα η πολιτική μας σε επιστημονικά στοιχεία και να μην κρύβει ποτέ ούτε τις επιφυλάξεις ούτε κάποιους συσταγμούς που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες. Εύσα έχει κάνει μια δουλειά εδώ και γνώρισε μεγάλη κριτική για τη μεροληψία της, για την έλλειψη καμιά φορά ανεξαρτησίας και ε, η κυρία Ρένκενς παραμένει ε, υπό αμφισβήτηση ακόμα και σήμερα. Έχω λοιπόν τις εξή ερωτήσεις. Θα δεσμευθείτε έτσι ώστε το πάνελ των γενετικά τροποποιημένων θα να αποφεύγει τις συγκρούσεις σεβόμενο ε, ε Κείμενε νομοθεσίε, τις διατάξει, τα επιστημονικά στοιχεία, όπως το Δεκέμβριο του 2008 συνέστησαν οι Υπουργοί των Κρατών Μελών στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντο. Ευχαριστώ. The basis of uh, our... Η βάση των αποφάσεων μα στον τομέα αυτό, όταν πρόκειται για προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε και οδηγίες που δίνουμε, στην υγεία και στην ασφάλεια των τροφίμων, είναι πάντα η επιστήμη. Πάντα η επιστημονική ενημέρωση καθοδηγεί τις συμβουλές μας. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, ιδιαίτερη σημασία να ε, γίνεται αυτό με σωστό τρόπο. Γιατί θα πρέπει πάντα η ενημέρωση να είναι απολύτως αντικειμενική και βάσει επιστημονικών στοιχείων. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα εξασφαλίσω με τις υπηρεσίες μου ε, όλες οι πληροφορίε και εκτιμήσεις που θα λαμβάνουμε να είναι. Θα είναι ανεξάρτητες για την παροχή συμβουλών μιλώ και θα μελετήσω τη δυνατότητα ή το ενδεχόμενο να θεσπίσουμε και τακτικούς ελέγχους και αναθεωρήσεις των θεμάτων ανεξαρτησίας των διαφόρων ε, υπηρεσιών ε, και οργανισμών, agencies. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντηση αυτή, αλλά οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αξιολογούνται από στοιχεία που δίνει η βιομηχανία η ίδια και δεν έχουν πρόσβαση ούτε οι ανεξάρτητοι επιστήμονες ούτε οι πολίτες παρά τα όσα αντίθετα ορίζονται. Και επίση μελέτε δείχνουν ότι χρειάζονται επιπλέον στοιχεία. Δεσμεύεστε να αναθέσετε σε ανεξάρτητου δημόσιου φορεί ε, τον έλεγχο και τη μελέτη αντικτύπου για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και να ε, έχουν πρόσβαση επιστήμονες στο γενετικό υλικό, όλα αυτά συνιστούν τμήμα της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση θα δίδεται σε όλους τους ε, ενδιαφερομένους και αφού διαβουλευόμαστε δημοκρατικά με όλους τους ενδιαφερμένους φωνείς, νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνεται αναθεώρηση ανεξάρτητη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν υπάρχει ε, κάποιο τέτοιο ζήτημα και πιστεύω ότι ο έλεγχος ε, αυτών των αποφάσεων επίσης θα ήταν κάτι το χρήσιμο. Σας παρακαλώ ε, να καταλάβετε ότι είναι θέματα αυτά για μένα που θα χρειαστεί να εντρυφήσω περισσότερο κατά τη διάρκεια της ε, εργασίας μου, των κατοικών μου σε περίπτωση που με δεχτείτε και μου αναθέσετε αυτό το χαρτοφυλάκιο, αλλά είμαι υπέρ ε, των ελέγχων και υπέρ της ενημέρωσης ε, για τις αποφάσεις βάσει των οποίων προχωρούμε σε άσκηση πολιτικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόπουλος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, χρειαζόμαστε σίγουρα πριν το καλοκαίρι μια αναθεωρημένη νομοθεσία σχετικά με τις μεταφορές ζώων. Επίσης, χρειαζόμαστε συγκεκριμένη νομοθεσία για να αποτρέψουμε στην ευρωπαϊκή αγορά τις τροφές που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. Τι θα κάνετε. Σχετικά με τα μεταλλαγμένα, που όπως βλέπετε απασχολεί εδώ το σώμα, ακριβώς επειδή υπάρχουν και οι εκτιμήσεις ότι η διάσπαση των αρμοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη διάθεση Υγείας έχει στόχο να μειώσει την ε, αποτελεσματική προστασία των πολιτών. Πώς θα διασφαλίσετε ότι όλες οι περιβαλλοντικές παράμετροι, ιδίω οι συνέπειες των γενετικά τροποποιημένων στη βιοπικιλότητα, αλλά και οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από την είσοδο στην αγορά των γενετικά τροποποιημένων πώς θα ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των κινδύνων. I Μάλλον συμφωνώ μαζί σας από τις πληροφορίες που είδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ότι υπάρχει κατακαιρματισμός στον τομέα και πιστεύω επίσης ότι η εισαγωγή του θέματος των ζωοτροφών από κλωνοποιημένα ζώα εντός της οδηγίας Novel Food μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα όχι μόνο για την ίδια τη συζήτηση για το θέμα της κλωνοποίησης αλλά και για τα άλλα θέματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν προς όφελος των πολιτών μας. Αυτό που θα συμβουλεύσω λοιπόν και του του να σας πω ότι είμαι εδώ μόνο μερικές εβδομάδες, μόλις τώρα ξεκινώ να αντιμετωπίζω αυτού του είδους τους φακέλους, δεν μπορώ εδώ να φανώ ως ειδήμων ότι έχω όλες τις λύσεις που αναμένουν όλοι, αλλά αυτό που θα μπορούσε να συμβεί κατά την άποψή μου είναι να υποβάλουμε ως πρόταση να γίνει μια ειδική αξιολόγηση για το θέμα της κλωνοποίησης και να υποβάλουμε μια έκθεση. Πιστεύω και το συζήτησα ήδη αυτό με τις υπηρεσίες μου. Πιστεύω ότι εντός ενός έτους μπορούμε να υποβάλουμε μια έκθεση για το θέμα της κλωνοποίησης που μετά μπορεί να συζητηθεί με εσάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, δεν θεωρώ ότι απαντήσατε για τα γενετικά τροποποιημένα και δεν παίρνετε υπόψη σας από ό,τι φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών είναι αντίθετη στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, πώς θα διασφαλίσετε το δικαίωμά τους να κάνουν ενημερωμένες επιλογές όταν πρόκειται για τρόφιμα που έχουν παραχθεί από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα αναλάβετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα και φυσικά ε, με το, ε, αυτό που ρώτησα πριν, για την, ε, να πάρετε υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και την βιοπικιλότητα. Και βέβαια οι πρωτοβουλίες αφορούν και την υποχρεωτική σήμανση των τροφίμων και σχετικά με την προέλευσή τους από ζώα που έχουν τραφεί από γενετικά τροποποιημένα. Κατανοώ ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για τέτοιου είδους θέματα και ότι υπάρχει μια κίνηση ή ένα αίτημα από ορισμένου, ακόμα και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, για σήμανση των ειδών διατροφής που προέρχονται από γάματα αφόμικρων. Αλλά αυτό που μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω είναι ότι ενεργά θα εξετάσω κάθε πτυχή του θέματος που είναι επιτάπητος, θα το συζητήσω στο κατάλληλο βήμα και βεβαίως θα συνεργαστώ και με εσάς εδώ στο κοινοβίλιο για αυτά τα διάφορα θέματα. Δεν πιστεύω ότι οι λύσεις αυτών των περίπλοκων θεμάτων είναι εύκολες πρέπει να δούμε όλες τις πτυχές διεθνής σχέσεις, ε, αφορά τη διατροφική ασφάλεια στο μέλλον, μπορεί να επηρεάζει λοιπόν πολλά θέματα και δεν νομίζω ότι η λύση μπορεί να βρεθεί από ένα και μόνο μυαλό. Πρέπει να είναι συλλογική μας προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. I was pleased to hear your opening remarks, uh, that Με χαρά είδα, κυρία Γιανακουδάκη, με χαρά είδα στα εισαγωγικά σας σχόλια ότι θα ασχοληθείτε με ασθενείς και καταναλωτές, αλλά βεβαίως αυτό δεν συνάδει με τα τελευταία σχόλιά σας να φύγει δηλαδή από το πακέτο η ενημέρωση των ασθενών. Μια και ο νέος Επίτροπος Υγείας θα είναι υπεύθυνο και για την ε, υπηρεσία για τα φάρμακα. Πώς θα εξασφαλίσετε την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη των ασθενών και τα οικονομικά συμφέροντα των γεωργών και την ουσιαστική έρευνα που απαιτείται για την Ευρώπη. Όπως είπα και αρχικά, πρώτα απ' όλα οι ασθενείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται ισχυρή δέσμευση για να είναι ανταγωνιστική και η γεωργία μας, γιατί τα συμφέροντα των ασθενών εξαρτώνται από μια ισχυρή και ανταγωνιστική γεωργία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα φάρμακα και τις περιθάλψεις που απαιτούνται από τους ασθενείς μας, εάν δεν έχουμε τις ροές κονδυλίων για τις απαραίτητες επενδύσεις για την έρευνα, εκμοντερνισμό και ανάπτυξη αυτών των νέων προϊόντων. Η υποστήριξη της φάρμα και τα συμφέροντα των ασθενών δεν είναι αντιφατικά αντιφατική στόχη μεταξύ της. Το γεγονός ότι είναι και μάλιστα σε ένα χαρτοφυλάκιο μας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε πολύ μεγαλύτερη συνέργεια ανάμεσα σε αυτά τα δύο θέματα. Πρέπει πάντως να τονίσουμε ότι θα πιέσουμε την φάρμα να προχωρήσει πολύ περισσότερο και θα έχουμε μία περιγραφή αρμοδιοτήτων η οποία βάζει τον ασθενή στο προσκήνιο αυτών των στόχων. Πιστεύω ότι η περίθαλψη των ασθενών είναι πολύ σημαντική με όλες τις, πτυχέ. πτυχές και νομίζω ότι έτσι θα συνεργαστούμε και με την φάρμα για να εξασφαλίσουμε ότι ο ασθενής θα ενημερώνεται και σωστά θα ενημερώνεται, δεν θα υποχρεώνεται να κάνει οτιδήποτε και αυτό θα σχετιστεί και με την ενημέρωση τους, του ασθενούς και ότι ο ασθενής θα ληφθεί σωστά υπόψη σε όλες τις πολιτικές που θα αναπτυχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρτίκα Λιωτάρ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Ντάλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει ξεχωριστή νομοθεσία για την κλωνοποίηση των, δο... των ζώων και το 2008 ήδη είχαμε ψήφισμα που ζητούσαμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα και να μην μπει καθόλου στην οδηγία για τα νέα τρόφιμα στο Novel Food. Και αν δεν υπάρξει ξεχωριστή πρόταση, είναι πολύ απίθανο να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Και αυτό σημαίνει ότι ένα πάρα πολύ ακαθόδε θέμα που αφορά την ασφάλεια ας πούμε, ε, των τροφίμων και την των τεχνολογία θα ε, είναι μετέωρο χωρί νομοθεσία. Ερώτηση. Συγκεκριμένα, πότε να περιμένουμε συγκεκριμένη πρόταση για τα κλωνοποιημένα ζώα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντηση. Όπως σας είπα και προηγουμένως, για το θέμα της κλωνοποίησης, ελπίζουμε εντός του έτους να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε έκθεση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της κλωνοποίησης. Όπως είπατε και έχετε απολύτως δίκιο. Χρειάζεται κάποια δράση, οπωσδήποτε γιατί η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να ε, παράγουμε και για τη βιομηχανία και για τους ασθενείς τους ίδιους και για την εσωτερική αγορά στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αγορά με μεγάλη ανασφάλεια. Αυτό που χρειάζεται είναι ασφάλεια. Τι σημαίνει όμως ασφάλεια. Σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να είμαστε σε θέση να κατανοούμε όλοι τις θέσεις ε, του καθενός και να προτείνουμε τις απαραίτητες λύσεις που θεωρούμε ότι είναι οι καλύτερες και οι πιο πρόσφορες και μακροπρόθεσμα για όλους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να το θεωρήσει κατάκτησή του ε, ότι θα ε, επιβάλλει τη γνώμη του και θα καρφώσει τη σημαία του. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον των καταναλωτών και είμαι προσιλωμένος προς την κατεύθυνση αυτή να συνεργαστούμε για να το επιτύχουμε. Εργάστηκα και θα εργαστώ ε, με τις υπηρεσίες μου πάρα πολύ στενά, όπως ήδη έχω εργαστεί για να ενημερωθώ και μαζί σας θα συνεργαστώ πάρα πολύ στα θέματα αυτά. τελειώνοντας την παρουσίασή μου, δεν πρόλαβα να σας πω αυτά που ήθελα, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με ορισμένους από εσά και εντυπωσιάστηκα από το βάθος των γνώσεών σας και ε, την εμπειρία σας. Και είναι λογικό, διότι εσείς φέρετε εδώ τις προσδοκίες ε, και ε, τις απόψεις των τοπικών φορέων. Ο στόχος είναι κοινός όμως, να αυξηθεί η ευημερία των λαών μας το Κοινοβούλιο εδώ θέλουμε ε, και εμείς μαζί σας να κάνουμε προτάσεις για λύσεις και γι' αυτό θα συνεργαστώ μαζί σας και είμαι πλήρως δεσμευμένος στην κατεύθυνση αυτή. Ναι, αυτό που με, μου απαντήσετε είναι για τους ασθενείς. Εγώ σας ρώτησα πότε θα φέρετε πρόταση συγκεκριμένη για την κλωνοποίηση των ζώων. Και η συμπροματική ερώτηση είναι εξή. Οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν θέλουν κλωνοποιημένο κρέας, πώς θα εξασφαλίσετε ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ε, δεν θα προταχθεί το ε, συμφέρον των βιομηχανιών, αλλά το συμφέρον των καταναλωτών και της υγείας του; Δεν μίλησα για ασθενείς, μίλησα για το τι θα κάνουμε εμείς. But... Uh, Μάλλον η διερμηνία αυτή λέει ο κ. Ντάλι. Αλλά εγώ σα είπα τι θα κάνουμε εμεί. Εμεί θα καταθέσουμε πρόταση για το θέμα αυτό τη κλωνοποίηση των ζώων. Αυτό σα είπα προηγουμένω. Και το τι θέλει ο κόσμος και τι θα γίνει με το εμπόριο. Και τη βιομηχανία και ε, τις απαιτήσει. Πρώτα ο κόσμος, πρώτα οι άνθρωποι, πρώτα οι καταναλωτές. Και εκείνου θα πρέπει να υπηρετούμε. Και δεν θα πρέπει να το φορτίσουμε συναισθηματικά. Θα πρέπει ε, αντικειμενικά και νυφάλαια να δούμε τι θέλουν οι πολίτες. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση κάποια αίσθηση που έχουμε ή, ή κάποιες ε, παραδοχές. Να ε, δούμε τι θέλει ο κόσμος. Ε, πιθανότατα θέλει αυτό που λέτε εσείς ακριβώς. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα ποια είναι και από εκεί και πέρα να αποφασίζουμε. Και η απόφαση είναι πάντα υπέρ των ε, ανθρώπων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω την εξή ερώτηση για την προστασία των καταναλωτών. Και μιλώ ιδιαίτερα για ουσίες που ε, διαταράσουν ε, τις ορμόνες, ακόμα και σε ελάχιστες ε, ποσότητες. Ποιες είναι οι ουσίες αυτές λοιπόν που διαταράσσουν τη σωστή λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος του οργανισμού. Τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να μην χρησιμοποιούνται και να μην κυκλοφορούν. Σε περίπτωση αμφιβολιών θα σταχθείτε υπέρ των καταναλωτών ή υπέρ της βιομηχανίας. και είστε βεβαίως ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ε, διατηρήσουν κάποιες επιπλέον απαιτήσει πέραν των όσων ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα απαγορεύοντας αυτές τις επιβλαβείς ουσίες. Για τη δημόσια υγεία επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να έχουν πιο αυστηρή νομοθεσία από την κοινοτική. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και εδώ οι βέλτιστες πρακτικές. Θα το κάνετε εσείς. I believe that, uh, Πιστεύω ότι απαγορεύεται να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κρέας από ζώα που έχουν ε, τραφεί με ορμόνες. Θα διατηρηθεί αυτή η πολιτική και αυτό εμείς θα ε, υπερασπιστούμε όσο μπορούμε και στεναρότατα και διεθνώς. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τις εθνικές νομοθεσίες και κατά πόσο επιτρέπουμε σε χώρες να έχουν υψηλότερες προδιαγραφές από την εναρμονισμένη ε, νομοθεσία, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εκτός αν με πείσετε περί του αντιθέτου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, λέγω, διότι αυτό θα είναι εις βάρος της εσωτερικής αγοράς. Η εσωτερική αγορά έχει ωφέλη για τον καταναλωτή. Η εσωτερική αγορά δεν ε, είναι προς το συμφέρον μόνο των οικονομικών ε, ε, φορέων, αλλά και των καταναλωτών. Και είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε και την εσωτερική αγορά στη διαδικασία λήψη των αποφασιών μας. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Εν τη αυτή περιπτώσει, Υπάρχουν κάποιες χώρες που θα δουν ε, την νομοθεσία τους να οπισθοδρομεί και να μειώνεται η προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τα σήμερα ισχύοντα προς αυτή την κατεύθυνση. Προσανατολίζεστε από ό,τι φαίνεται. Μάλλον. Διότι Πώς θα γίνει να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν όλες οι χώρες να είναι στο ίδιο επίπεδο. Κάποιες είναι ήδη πιο προηγμένες. Γι' αυτό σας ρώτησα για τις βέλτιστες πρακτικές. Εγώ θα πιέσω να υπάρχει παντού υψηλή προστασία. Το θέμα είναι προστασία ναι ή όχι. Για θέματα υγείας το ζήτημα είναι το σωστό επίπεδο προστασίας που θα πρέπει να επιμείνουμε να απολαμβάνουν οι πολίτες μας υπάρχει ένα σωστό επίπεδο προστασίας, το οποίο θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να προστατεύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει παντού να ισχύει η ισότητα. Ε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά και διπλές προδιαγραφές στη δημόσια υγεία. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι υποστηρικτής αυτού του φαινομένου ε, δύο ταχυτήτων προστασία και στο θέμα αυτό και αλλού θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το επίπεδο των προδιαγραφών μας και το προτύπο μας είναι το σωστό και θα βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Ερχόμαστε στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων με την κυρία Ζόμπερ. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές. Αυτό ισχύει και για την διατροφή. Έχει το δικαίωμα να έχει και σαφή, ξεκάθαρη πληροφόρηση για τα προϊόντα που καταναλώνει. Όμως, όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προχωρεί σε εκπαίδευση του καταναλωτού με απαγορεύσεις διαφημίσεων, με αρνητική παρουσίαση ε, σε ετικέτες και ούτω καθεξής, πάνε να βάλουν Ζουρνομανδία στον καταναλωτή, ώστε και καλά να είναι υγιής. Δηλαδή δεν ξέρει πια ο πολίτης τι πρέπει να διαλέξει και θα του επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, συχνά λείπει η επιστημονική θεμελίωση από ε, τις εκθέσεις των γενικών διευθύνσεων. Για πολιτικούς λόγους υιοθετούνται κάποιες τιμές ή κάποια όρια χωρίς απαραίτητα επιστημονική θεμελίωση. Μπορείτε να βεβαιώσετε ότι θα φροντίσετε αυτό να αλλάξει. Απάντηση. Δεν μπόρεσα να ακούσω μέχρι τέλους, λόγω του ότι διακόπη μετάφραση, την δεύτερη ερώτησή σας. Πάντως για την πρώτη ερώτηση, πιστεύω και πάντως η γνώμη μου είναι η εξής. Δεν θα ήθελα να πω στον Ευρωπαίο πολίτη τι να τρώει. Αλλά θέλω να τους πω τι είναι αυτό που τρώνε. Ε, περί αυτού πρόκειται. Ολόκληρη ιστορία αυτή είναι. Εκεί πραγματικά πρέπει να πιέσουμε να πιέσουμε έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα, τις ικανότητες στον πολίτη, στους πολίτες για να μπορούν να διαλέξουν εφόσον βέβαια διαθέτουν την επαρκή πληροφόρηση. Τώρα πόση πληροφορία θα βάλουμε πάνω σε μια ετικετούλα μιας καραμέλας, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί ίσως ε, ε, κάποια στιγμή πάει και πολύ. Πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς τη λογική. Όμως ο στόχος είναι ο καταναλωτής πρέπει να είναι ενήμερος. Αυτό είναι ουσιώδες. Διότι αλλιώς τι απόφαση μπορεί να λάβει εάν δεν γνωρίζει όχι ότι κάτι είναι καλό ή κακό για την υγεία του. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει και καλά να πούμε στον κόσμο τι είναι καλό για την υγεία του. Να αποφασίζουν μόνοι του οι άνθρωποι τι είναι καλό και τι είναι καλό για την υγεία του. Όμω, πρέπει να του λέμε τι τρώνε, τι περιλαμβάνουν τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουν, ώστε οι ίδιοι να μπορούν εν τέλει να αποφασίζουν. Πιστεύω λοιπόν ότι η ικανότητα αυτή που μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή είναι και παραπέρα από αυτό. Δηλαδή οι καταναλωτές είναι μια στρατιά ολόκληρη ανθρώπων οι οποίοι με τις αποφάσεις τους κατευθύνουν τις αγορές. Ανά πάσα στιγμή ε, λαμβάνονται εκατομμύρια αποφάσεις στις αγορές. Και εγώ θέλω οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι για το τι καταναλώνουν, ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορούν να επηρεάζουν και την κλιματική αλλαγή και την ευημερία των ζώων και όλες τις άλλες πολιτικές τις οποίες ασκούμε είπαμε να ασκήσουμε η ε, Συμπληρωματική ερώτηση, η δεύτερη, σας ευχαριστώ για την πρώτη απάντηση. Συχνά η επιστημονική θεμελίωση λείπει από τις εκθέσεις της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, Προστασίας Καταναλωτών. Για παράδειγμα, για την θρεπτική αξία. Και εγώ ισχυρίζομαι ότι συχνά είναι πολιτικοί οι λόγοι όταν δηλαδή πολιτικά κάτι θέλουν να επιτύχουν για να οθήσουν τους καταναλωτές σε ένα υγιή τρόπο ζωής. Και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία επιστημονική θεμελίωση για τα θέματα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας. Είναι σωστό για πολιτικούς λόγους να καθορίζονται τιμές κατόφλια ακόμα και αν η επιστήμη λέει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν και δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική θεμελίωση. απάντηση. Εδώ θα προβώ σε δήλωση. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι η μακροπρόθεσμη ευημερία του Ευρωπαίου πολίτη. Κάθε απόφαση που θα λάβω θα πρέπει να βασίζεται σε αυτή τη λογική. Θα υπάρχουν και άλλα συμφέροντα και περιφερειακά συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό λόγο σε ό,τι με αφορά. Καθένας θα πρέπει να παίξει το ρόλο του στον διάλογο. Βεβαίω πρέπει να ακουστούν όλε οι πλευρέ, όλα τα συμφέροντα και πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν θα λάβουμε μια τελική απόφαση. Αλλά ο τελικό γνώμονα πρέπει να είναι οι σωστέ προτεραιότητε. Και οι δικέ μου προτεραιότητε, και το δηλώνω και θα το δηλώσω αυτό μέχρι ναυτία. Η δική μου προτεραιότητα είναι η μακροπρόθεσμη ευημερία του Ευρωπαίου πολίτη. Σα ευχαριστώ, κύριε Ροτ Μπέρεντ. Κύριε Νταλή, οι χώρες μέλη έχουν περιορισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή επιρροή σε θέματα πολιτικής. Υπάρχει και αντίσταση στην προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την πολιτική υγείας, κυρίως για την υγιεινή των τροφίμων, την ε, επιτήρηση και την, την εποπτεία της χρήσης των φαρμάκων κλπ. Εσείς κύριε Νταλή θα Προσπαθήστε να επιτύχετε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας αντιστεκόμενος ή ε, αντιπαρατηθέμενος στην αδράνεια του Συμβουλίου και θα ασκήσετε την επιρροή σας ως ε, πρώην ε, Υπουργός Υγείας. Και ήταν, ποιος ήταν ο ρόλος σας στο Συμβούλιο όταν ήσασταν Υπουργός Υγείας και επομένως συμμετείχατε σε αυτό το όργανο. απάντηση. Στην σταδιοδρομία μου αναμίχθηκα βέβαια στην εκπόνηση πολλών νομοθετημάτων και, ε, και πρότεινα στο Κοινοβούλιο συχνά νομοσχέδια. Όμως ένα νομοσχέδιο δεν αξίζει ούτε καν το χαρτί που είναι γραμμένο εάν δεν περιλαμβάνει και τα περί της επιβολής του. Η επιβολή και να πω και κάτι άλλο. Όταν κάποιος προτείνει κάποιο νομοθέτημα, πρέπει να είναι ορατό το στοιχείο της επιβολής. Πώς θα επιβληθεί η σχετική νομοθεσία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντάτε ακόμη και στη μελέτη επιπτώσεων της νομοθεσίας. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Είναι δυνατόν να επιβληθεί. Είμαστε επαρκώς οργανωμένοι ώστε να φροντίσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας. Διότι αλλιώ θα έρθετε θα μου πείτε, μα δεν συμμορφώνονται οι χώρε μέλη. Πρέπει λοιπόν να τα επιβάλλουμε τα πράγματα αυτά. Και πρωτίστω οφείλουμε να ενισχύσουμε τι διαδικασίε επιβολή και την ικανότητα επιβολή. Από την άλλη μεριά, καλούμαστε να συνεργαστούμε με τι χώρε μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά του έχουν όντω την ικανότητα να επιβάλλουν. Και τώρα ε, σας τα λέω αυτά γνωρίζοντας και την άλλη πλευρά της ιστορίας και μπορώ να σας καταστήσω κοινωνούς του πώς, ποια είναι η νοοτροπία της άλλης πλευράς. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ικανότητα επιβολής των ίδιων χωρών μελών. Ορισμένες φορές ε, θέλουν ή και μπορεί να μην θέλουν να συμμορφωθούν σε κάποια, σε κάποια νομοθεσία. Όμως πρόκειται και για προτεραιότητες που οφείλουμε να πείσουμε τις χώρες ότι πρέπει να τις σεβαστούν και κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους και τις ικανότητες που οφείλουν να αναπτύξουν για να μπορέσουν να επιβάλλουν. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ, ναι, συμφωνώ με την επιβολή, αλλά νομίζω ότι βιαστήκατε λιγάκι. Θα μιλήσουμε για επιβολή όταν θα έχουμε ήδη την νομοθεσία. Το δικό μου παράπονο είναι ότι οι χώρες μέλη δεν συμφωνούν σε μια ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέλουν να την μπλοκάρουν, να την αποδυναμώσουν. Θα είστε ισχυρός επίτροπος ώστε να τις αναγκάσετε τις χώρες να τις σπρώξετε, να του δώσετε μια κλωτσιά αν χρειαστεί για να πάρουν μπρος και να κάνουν αυτά που πρέπει. Δικό σας είναι το καθήκον αυτό. Πόσο ισχυρός θα εμφανιστείτε. Θα είμαι ισχυρός. Πιστεύω ότι αν εξετάσετε το παρελθόν μου και τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκα στην ίδια μου την πατρίδα θα δείτε ότι μπορώ να δείξω δύναμη. Καμιά φορά μάλιστα με επέκριναν επειδή ήμουν υπερβολικά ισχυρό και αυστηρό στην πρόθεση κάποιων νομοθετικών επιλογών. Αλλά όταν κάνουμε κάτι που αξίζει τον κόπο, και εγώ δεν θα κάνω τίποτα που να μην αξίζει τον κόπο, θεωρώ, πιστεύω, ότι πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και τότε θα αφιερώσω όλη μου την ενέργεια στην επιτυχία της απόπειρας αυτής. Η ισχυρή επιτροπή, ισχυρή επίτροπη. Αυτό θέλουμε και εμείς. Η κυρία Μπίλτ Με χαρά άκουσα την ισχυρή σας δέσμευση για να δοθεί μεγάλη εξουσία στους καταναλωτές και χαίρομαι που θα αντισταθείτε στα κράτη-μέλη. Έχω δύο ερωτήσεις για την σήμανση των ειδών διατηροφής που τώρα συζητούμε. Πώς θα συμφιλιώσετε την ανάγκη να υπάρχει απλή και σωστή ενημέρωση και τις Ανησυχίε των βιομηχανιών, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ότι είναι υψηλότερο το κόστος για αυτού. Μπορούν να κερδίσουν και οι δύο. Και πώς και σε ποιο επίπεδο εναρμόνισης θεωρείται ότι πρέπει να φτάσουμε. Μετά το κεφάλαιο 6 και 7 τη υφιστάμενη πρόταση για εθνικές διατάξεις, υποχρεωτικές εθνικές διατάξει και εθελοντικά ε, εθνικά προγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένας τρόπος κατακαιρματισμού της αγοράς, σύγχυσης του καταναλωτού, παρεμπόδισης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πώς θα αντισταθείτε στα κράτη-μέλη για να περιορίσετε ότι οι εθνικές διατάξεις δεν θα στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. I Κατανοώ τα θέματα των διαφόρων απαιτήσεων που επιβάλλουμε στους κατασκευαστές μας και στους εμπορευόμενους για να πληρούν τις απαιτήσει για ενημέρωση των καταναλωτών. Είναι σημαντική η ενημέρωση των καταναλωτών και αυτή πρέπει να τη σεβαστούμε στις αποφάσεις μας. Στα πλαίσια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν διατάξεις ευελιξίας ήδη εντός της πληθώρας νομοθετικών κειμένων που διαθέτουμε και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε γιατί δεν είναι συμφέρον μας να προωθήσουμε πολιτικές που θα είναι επιζήμιες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των οικονομιών μας. Πρέπει όμως επίσης να σεβαστούμε και τα πρότυπα ενημέρωσης των καταναλωτών και σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη και τα εθελοντικά εθνικά προγράμματα και την διαφορά που θα υπάρχει στις διάφορες αγοράς, επαναλαμβάνω τα όσα είπα προηγουμένως, ότι νομίζω ότι θα πρέπει όσο το δυνατόν να μειώσουμε τις διαφορές στην εσωτερική αγορά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει κανένας να προχωρήσει με μικρότερους, με αργότερους ρυθμούς για να επιτύχει τους στόχους τους και όχι να υπάρχει μία και γρήγορη λύση για μία συγκεκριμένη πρόταση. Και η εμπειρία μου μου δείχνει ότι μία σταδιακή προσέγγιση μερικές φορές είναι πιο επιτυχής και πιο γρήγορη και μπορεί πολλές φορές αυτή να είναι η προσέγγιση που θα υιοθετήσουμε. Έχουμε ένα τελικό στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε, αλλά το να τους πείσουμε τελικά ότι είναι προς όφελος όλων, αυτό είναι το σημαντικό. Σας ευχαριστώ για την ισορροπημένη σας απάντηση. Άλλο αμφιλεγόμενο θέμα είναι η σήμανση για την χώρα προέλευσης. Δείχνουν οι έρευνες ότι ο κόσμος θέλει χνηλασιμότητα αλλά για την βιομηχανία αυτό είναι επιπλέον κόστος και όχι θέμα προστατευτικού. Είστε υπέρ της υποχρεωτικής σήμανσης για την χώρα προέλεσης για τα προϊόντα των ειδών διατροφής. Θεωρώ ότι η παρούσα κατάσταση είναι ότι η σήμανση της χώρας προέλευσης με εξαίρεση κρέας ψάρια είναι εθελοντικού χαρακτήρα με εξαίρεση εάν υπάρχει δυνατότητα παραπλάνησης του καταναλωτή. Τότε είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται και η χώρα προέλευσης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να παρεκκλίνουμε της κατάστασης αυτής αλλά όπως και όλα τα άλλα θέματα θα προχωρήσουμε σε αυτά τα πέντε χρόνια και πέντε χρόνια είναι πολλής χρόνος για να κάνουμε πολλές προσπάθειες και ελπίζω να κάνουμε προσπάθειες από κοινού και για αυτό και για άλλα θέματα. Αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από την ιεράρχηση που θα κάνουμε για το πρόγραμμά μας και το ποιους στόχους πρέπει να επιδιώξουμε για τους πολίτες μας και έτσι θα προωθήσουμε και το θέμα αυτό. Η κυρία Κέμπχαρτ. Ευχαριστώ. Κύριε Νταλή, θα είστε αρμόδιος και για εμπορεύματα και υπηρεσίες και εν προκειμένου η διασύνδεση κοινωνικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων καταναλωτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς και Καταναλωτών ανησυχούμε, ανησυχούμε πολύ όχι επειδή εσεί είστε ο υποψήφιο επίτροπος, αλλά διότι διαπιστώνουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε αυτό το τομέα των ε, υπηρεσιών. Δεν είναι μόνο η κυρία Ρέντινγκ, η κυρία Κρούς, είναι και ο κύριο Μπαρνιέ και ο κύριο Ταζάνη. Και ε, όλοι αυτοί είναι συναρμόδιοι. Εμείς ανησυχούμε. Πώ μπορεί να εξασφαλιστεί η συνοχή στην προστασία των καταναλωτών για εμπορεύματα και υπηρεσίε. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα, πως έχετε οργανωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσετε αυτή τη συνοχή στην ε, ε, προστασία του καταναλωτού σε θέματα εμπορευμάτων και υπηρεσιών και ποιος είναι αρμόδιος εν τέλει για το συντονισμό. Είμαι ο Επίτροπος Αρμόδιος για όλα τα θέματα προστασίας καταναλωτών μέσα στο Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων και γι' αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε όλες οι συζητήσεις στο Συμβούλιο να περιλαμβάνουν και μια πτυχή προστασίας του καταναλωτού. Όταν λέμε κατακαιρματισμό, πράγματι, όλα όσα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν σχέση με τους ανθρώπους. Επομένως κάθε χαρτοφυλάκιο στην πραγματικότητα έχει και μια πτυχή προστασίας καταναλωτού. Εγώ θα φροντίσω ώστε κάθε πρόταση που θα υποβάλλεται στο συλλογικό σώμα των επιτρόπων θα έχει θα λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και τις σχετικές ιδέες και σκέψεις. Εγώ θα θεωρώ εαυτόν θεματοφύλακα της προστασίας των καταναλωτών. Είναι αληθές ότι υπάρχουν πολλοί τομείς όπου ε, ο καταναλωτής έχει ε, υψηλό προφίλ, για παράδειγμα, στην ενιαία αγορά, σε θέματα επικοινωνίας κλπ. Της κυρίας Ρέντινγκ επίσης που και εκεί συμμετέχει στην ομοθεσία προστασία του καταναλωτού και αυτό είναι καλό γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ώστε η οπτική αυτή της προστασίας του καταναλωτού ε, θα είναι ανάγλυφα ε, παρούσα διαρκώς. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Και όσο θα συντονίζουμε εμείς αυτές τις απόψεις, δεν ανησυχώ. Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο από τον οποίο θα εργαστούμε και θα συνεργαστούμε, αλλά πάντως αναλαμβάνω την δέσμευση να είμαι ιδιαίτερα επιμελής ε, σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτού του συντονισμού. Και βεβαίως ε, θα επανέρχομαι εδώ να σας βλέπω συχνά και αν δεν κάνω καλά τη δουλειά μου θα περιμένω από εσά να μου το πείτε. Να μου πείτε πού χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις. η κυρία Γκέπχαρτ πάλι. Άκουσα ευχαρίστω τα όσα είπατε και ελπίζω όντω να υλοποιηθούν. Υποβάλλω μια ακόμη ερώτηση την οποία είχαμε κάνει και με συμφωνία με τον κύριο Μπαρόσο, γιατί και προ δύο ημερών στην ακρόαση της κυρίας Ρέντινγκ προκλήθηκε η εντύπωση ότι η ίδια θα έκανε τον συντονισμό. Ήθελα λοιπόν να είμαι βεβαία ότι εσείς θα αναλάβετε τον συντονισμό Τη υπόθεση τη υποστασία του καταναλωτού. Απάντηση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτά που λέω εδώ απηχούν τις συζητήσεις που έκανα με τον πρόεδρο Μπαρόσο και αυτά μου είπε εξηγώντα μου τις διάφορες πτυχές του χαρτοφυλακίου μου. Ο κύριος Λέχνερ κύριε υποψήφια επίτροπε. Συχνά ακούσαμε περί προστασίας καταναλωτού και κυρίως τον έλεγχο, την ε, παραχώρηση δικαιωμάτων στον καταναλωτή κτλ. Όμως από την άλλη πλευρά τώρα, τι σημασία έχει ο ανταγωνισμός από τη δική σας σκοπιά. Πώς εξυπηρετεί δηλαδή την προστασία του καταναλωτού και επομένως και την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και ότι ο καταναλωτής δεν θα στρέφεται αυτομάτως στο φθηνότερο προϊόν αλλά θα εξετάζει και θα λαμβάνει υπόψη και την ποιότητα και πώς επίσης θα λαμβάνονται υπόψη διάφορες διαφορετικές παραδόσεις και επομένως η αρχή της επικουρικότητας στην υπόθεση αυτή της προστασίας του καταναλωτού και κατά πόσον εσείς θέλετε να επιβάλλετε πάντοτε μια συνολική επισκόπηση κόστους και ωφέλους. Γιατί εν τέλει ο καταναλωτής ανάλογα και με τις ε, αποφάσεις του μπορεί να πληρώνει το κόστος αργότερα. Όταν μιλούμε για ανταγωνισμό και όπως σωστά είπατε, είναι θέμα τιμής και ποιότητας. Στο σύστημά μας και όπως αυτό έχει λειτουργήσει ως τώρα και ελπίζω θα μπορέσουμε να το ενισχύσουμε κιόλα, το θέμα της ποιότητας έχει ουδετεροποιηθεί, διότι έχουμε εξασφαλίσει ώστε κάθε τι που μπαίνει στην αγορά μας υπακούει σε κάποια κριτήρια ποιότητας. Αφήστε λοιπόν έχει ουδετεροποιηθεί το θέμα αυτό, σημαίνει ότι όσα ε, καταναλώνουμε και αγοράζουμε δεν είναι επικίνδυνα, είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια ποιότητας. Νομίζω ότι οι άλλες σκέψεις θα είναι πιο σημαντικές πια. Βεβαίως Υπάρχει ποιότητα και υπάρχει άλλη ποιότητα. Υπάρχει λοιπόν η ελάχιστη ποιότητα και υπάρχει κάτι άλλο που είναι καλύτερο σε ποιότητα. Αλλά εν τέλει η ελεύθερη επιλογή του καταναλωτού θα είναι και εκεί βρίσκεται η ομορφιά της ενιαίας αγοράς. Ότι ο καταναλωτής θα έχει μπροστά του ένα ολόκληρο φάσμα προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα σε αυτόν. Ένα ολόκληρο φάσμα διαφόρων επιπέδων ποιοτικών αγαθών σε διαφορετικές τιμές που μπορεί να ε, ε, αγοράσει παίρνοντα τα από το ράφι. Και η δική του απόφαση θα είναι βεβαίω αυτή που θα κρίνει εν τέλει. Τρίτος γύρος, η κυρία Ρατβιλέ Μορκουνάιτε. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου ερώτηση έχει σχέση με την οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών και την κινητικότητα τη διασυνοριακή των ασθενών. Για μένα είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα αυτό. Η οδηγία θα είναι πολύ χρήσιμη κατά την απόψή μου, διότι ένα από τα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές είναι η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Η οδηγία αυτή λοιπόν θα είναι καλό παράδειγμα για τους πολίτες της Ένωσης. Θα δείξει δηλαδή τους πολίτες της Ένωσης πώς η Ένωση ίδια επηρεάζει την καθημερινή του ζωή. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να είστε πιο δραστήριο στην αναζήτηση κοινή θέση στα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει εργαστεί πολύ ε, για την οδηγία αυτή. και η έκθεση του Κοινοβουλίου ε, έστειλε ένα θετικό πολιτικό μήνυμα για τις ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτει. και πόσο ε, αναγκαία είναι η οδηγία. Η κυρία Κροστέτ μάλιστα ήταν πάρα πολύ δραστήρια και θα ήθελα να την ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος εδώ και να αποτίσω ένα φορτιμής. Προτίθεστε να επανέλθετε λοιπόν, ε, να επαναφέρετε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, στην πολιτική σας ατζέντα, το πρόγραμμά σας και πώς δεσμεύεστε προς την κατεύθυνση αυτή. Και εγώ πιστεύω, όπως και εσείς, ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να προωθηθεί, να προχωρήσει. Γνωρίζουμε όλοι τι συζητήσεις προηγήθηκαν στο Συμβούλιο και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Και η προκάτοχός μου έκανε πάρα πολλές προσπάθειες για να εξασφαλίσει ε, την πρόοδο σε αυτό το θέμα. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια συμφωνία και μια αποτελεσματική τέλη πολιτική για τα δικαιώματα και την κινητικότητα των ασθενών. Μαθαίνω ότι η Ισπανική Προεδρία δήλωσε προθυμία, ε, το προωθεί πάρα πολύ το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της, δηλώνει, και η πρώτη δράση μου ουσιαστικά, σε περίπτωση που με εγκρίνεται, θα είναι να μεταβώ και να έχω μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας ε, στην Ισπανία. Να μεταβώ στη Μαδρίτη δηλαδή και να μιλήσω με τον αρμόδιο Υπουργό για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου ε, στο θέμα αυτό και να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Ελπίζω, δεν έχω και ελπίζω το θέμα αυτό να λυθεί το συντομότερο. Ευχαριστώ. Η Γκλένις Βίλμοντ. Ε, κύριε Υποψήφια Επιτρόπη, χαίρομαι για το γεγονός ότι έχει πάει στη δημόσια υγεία και έχει φύγει από τη βιομηχανία το θέμα των φαρμάκων. Είναι σημαντικότατο εδώ το θέμα της δημόσιας υγείας και όχι ε, το θέμα της βιομηχανίας όταν μιλάμε για μια φαρμακολογική πολιτική. Είστε βέβαιος όμως ότι η φαρμακοβιομηχανία βγάζει φάρμακα καλά και υγιή που ε, θα αντιμετωπίζουν ε, νοσήματα που απειλούν τη ζωή των ασθενών και πώς θα είναι αρκετά προσιτά και προσβάσιμα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και φθηνά τα φάρμακα. Εδώ θίξατε τρία θέματα κλειδιά. Η ε, ύπαρξη των φαρμάκων, η πρόσβαση στα φάρμακα για όλους τους ενδιαφερομένους και η τιμή που βεβαίως ε, για να υπάρχει πρόσβαση στα φάρμακα θα πρέπει να είναι και η τιμή τους προσιτή. Κοιτάξτε, με τα φάρμακα στο χαρτοφυλάκι αυτό έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε τις αδικίες, τις ανισότητες, να έχουμε καλά φάρμακα ε, προσβάσιμα ε, προς όλους. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει και η φαρμακοβιομηχανία και εμείς να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να συναντηθούμε και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εντάξει, όλοι πολιτικοί είμαστε εδώ και ξέρουμε ότι τέτοιου είδους συνεννοήσεις δεν είναι θέμα να κάνει ο ένας για χάρη σε κάποιον άλλον. Πάντα εδώ πρόκειται για πώς να το πω, μια συνεννόηση που βασίζεται ε, στην συνειδητοποίηση ότι σε τελική ανάλυση έχουμε όλοι να κερδίσουμε από αυτό και το πιστεύω. Ε, θα πρέπει να πείσουμε τη φαρμακοβιομηχανία ότι και για εκείνους είναι καλή μια τέτοια λύση και να μας βοηθήσει να φτάσουμε στους στόχους μας τότε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή. Ευχαριστώ για την απάντηση αυτή. Γίνεται μεγάλη πίεση όμως ε, προς όλους μας από την φαρμακοβιομηχανία και το έχουμε όλοι ζήσει. Πώς ε, θα εξασφαλίσετε εσείς, τι προτίθετε να κάνετε για να προέχουν τα συμφέροντα και η φωνή των ασθενών. Ε, πρώτα απ' όλα επαφίομαι σε εσά, τους βουλευτές. Για να εξασφαλίσετε πέρα από το λόμπι και την πίεση που σας ασκούν προωθείτε εσείς τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των ασθενών που είναι και ε, οι ψηφοφόροι σας. Σας είπα, ε, θα συνεργαστώ μαζί σας και τι εννοώ. Είμαι πραγματικά ακράδαντα πεπισμένος ότι από εσάς θα ε, ε, παίρνω, θα δέχομαι ε, τα σχόλια και τις αντιδράσεις των πολιτών, όχι της φαρμακοβιομηχανίας. Η φαρμακοβιομηχανία δεν σας χρειάζεται εσά για να γίνει η φωνή της ακουστή. Έχει τη δική της φωνή. Εσείς είστε με την πλευρά των πολιτών σε ό,τι με αφορά και στις δικές μου λοιπόν διαβουλεύσεις και συζητήσεις έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το ρόλο του Κοινοβουλίου. Βεβαίως θα πρέπει να συνεννοούμαστε και να διαβουλευόμαστε και με τις οργανώσεις των ασθενών ε, για να μας λένε τα σχόλια τους. Ευχαριστώ. Από τη Μάλτα η επόμενη ερώτηση, ο Λουίς Κρέχα. Κύριε Ντάλι, σε μία από τις γραπτές σας απαντήσεις για τους μηχανισμούς διόρθωσης είπατε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαβούλευση για πιο αποτελεσματική λύση. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη και ένα παράδειγμα ήταν τα όσα συνέβησαν στην Μάλτα για τον ΦΠΑ για την ταξινόμηση αυτοκινήτων. Τώρα έχω την εντύπωση ότι είστε υπέρ ότι η Ένωση πρέπει να υιοθετήσει ε, λόγους για συλλογική διόρθωση και θα υπάρξει πρόταση το ταχύτερο δυνατόν έχοντας κατά νου ότι το θέμα αυτό είναι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια. of moving forward with collective ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό αποζημίωσης και διόρθωση των ζημιών για τους καταναλωτές. Η Γενική Διεύθυνση ΑΝΚΟ εργάζεται σκληρά για το θέμα αυτό και ήδη έχουν περατώσει μία μελέτη αντικτύπου για προτάσεις που θα υποβληθούν και έχουν περάσει ήδη από την Επιτροπή αξιολόγησης η οποία υπέβαλε κάποια σχόλια τα οποία η ΣΑΝΚΟ αυτή τη στιγμή εξετάζει. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει η βούληση και όχι μόνο η βούληση, ήδη η κίνηση για να υπάρχει τέτοιου είδους λύση. Όπως ξέρετε όμως, η άλλη μια διαδικασία για συλλογικές αγωγές και ε, αποζημιώσεις την επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην καταλήξουμε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση με αυτά τα δύο νομοθετικά κείμενα. Πιστεύω ότι χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος για να εξασφαλίσουμε ότι συντονίζουμε τις δράσεις μας πρέπει να εδώ να συνεργαστούμε και με την κυρία Ρέντινγκ για να έχουμε την βέλτιστη δυνατή νομοθεσία και μετά να προχωρήσουμε. Πιστεύω όμω επίσης ότι και ο καταναλωτής, γιατί στην ουσία εδώ μιλάμε για νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή και στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μιλάνε για προστασία του καταναλωτού από παραπλανητικό εμπόριο. Πιστεύω όμως ότι οι έννοιες είναι λίγο διαφορετικές και ότι στο τέλος θα πρέπει να έχουν συγκερασμένες προτα... προσεγγίσεις. Στην ίδια απάντηση είπατε ότι για να έχει εξουσία ο πολίτης πρέπει να έχει περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνούμε απολύτως με αυτό. Ποιες πρωτοβουλίες όμως θα λάβετε για να εξασφαλίσετε ότι οι πολίτες έχουν πληροφορίες που δεν είναι παραπλανητικές και δεν είναι διαφημίσεις. Επίσης, είπατε ότι η προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων είναι το αντικείμενο της πολιτικής μας. Ποια θα είναι η πολιτική σας ως Επιτρόπου για να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές. Απάντηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σήμερα εργαζόμαστε σκληρά, η Κομισιόν εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσουμε ότι η ενημέρωση που χορηγείται στον καταναλωτή είναι η σωστή ενημέρωση. Παραδείγματος χάρη, η πρωτοβουλία που αναλάβαμε για τις αξιώσεις σε θέματα υγείας. Αυτό αποδεικνύει. Δηλαδή, αν κάποιος παραγωγός υπερισχύει ότι το προϊόν του σας κάνει καλό, σας κάνει πιο αδύνατο, πιο ψηλό. Μπορεί να σας κάνει να αδυνατίσετε. Όλες αυτές, οι, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ελέγχονται και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι σωστές. Σωστοί όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Όμως ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο νομίζαμε. Και θα σας απαντήσω λίγαν συντόμως. Ευχαριστώ κυρία Σουζάνα Ρόιτοβα. Καλό απόγευμα κύριε Ντάλη, εδώ είμαι. Καλώ ήρθατε. Τα ερωτήματά μου αφορούν την προστασία των παιδιών από τα επικίνδυνα προϊόντα που έχουν εισβάλλει στην αγορά μας. Συνεργάζομαι με εμπειρογνώμονες για τα ελάχιστα πρότυπα που είναι απαραίτητα για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και εισαγωγής εισαγωγή, ασιατικών προϊόντων. Έχουμε πρότυπα για το σχήμα των αγκουριών, αλλά δεν έχουμε ορθοπαιδικά πρότυπα για τα παπούτσια των παιδιών. Είστε διατεθειμένος κύριε Επίτροπε να εισαγάγετε νομοθεσία για ελάχιστα πρότυπα για τα παπούτσια των μικρών και λίγο μεγαλύτερων παιδιών γιατί αυτού του είδους τα προϊόντα δημιουργούν μεγάλες ζημίες και πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε την προστασία των παιδιών σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Απάντηση. Ένα από τα ευάλωτα τμήματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι τα παιδιά. Και γι' αυτό τους προσδίδω ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να τα προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την εκμετάλλευσή τους. Ούτε μικρή ούτε μεγάλη εκμετάλλευση. Ούτε καν προωθώντας τους για προϊόντα που τελικά τους είναι επιζήμια. Έχουμε πρότυπα στην Ευρώπη και από ό,τι ξέρω κάθε πρότυπο που έχουμε στην Ευρώπη ισχύει και για όλα τα προϊόντα που εισαγάγονται από τρίτες χώρες. Τα πρότυπα λοιπόν που έχουμε ως κανόνας ισχύουν ισότιμα και σε ό,τι εισαγάγουμε. Αν τώρα υπάρχουν πρότυπα για παπούτσια ή για παιχνίδια. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή συζητούνται για να καταλήξουμε στα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται. Θα προσπαθήσω πάντως να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε τα κατάλληλα πρότυπα για να προστατεύσουμε όλα τα προϊόντα, αλλά ιδιαίτερα τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε πρότυπα που ισχύουν για παιχνίδια, αλλά όχι για τα παπούτσια των παιδιών. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας για το θέμα αυτό. Η απάντηση είναι ναι, αυτό θα κάνω, θα συνεργαστώ μαζί σας για αυτό το θέμα και άλλα θέματα για να εξασφαλίσω όλοι ότι τα προϊόντα που φτάνουν στα παιδιά μας είναι ασφαλή. Σαφέστατο είναι αυτό και ευπρόσδεκτο. Ο Τόιν Μάντερς, επόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Κύριε Ντάλι, καμιά φορά εμεί, οι πολιτικοί υπεραντιδρούμε στην προστασία των καταναλωτών και αυτό μπορεί να οδηγεί σε πολύ μεγάλη ε, πληθώρα πληροφοριών και γραφειοκρατικό φόρτο. Τώρα ο κύριο Μπαρόσο θέλει κατά 25% να μειώσει αυτό το γραφειοκρατικό φόρτο. Για να δίνεται αυτή η πληροφόρηση, εγώ προτιμώ το διαδίκτυο και μια ιστοσελίδα που να υπάρχει και ένας αριθμός αναφοράς για το προϊόν και αυτό κάνει τη ζωή όλων πιο εύκολη. Για παράδειγμα, στην κλωστοϊφαντουργία αλλά και στα τρόφιμα, κοιτάξτε αυτό το μπουκαλάκι πόσες πληροφορίες έχει τυπωμένες επάνω του το νερό ε, κατακλείζεται με πληροφορία το ε, προϊόν και είναι πληροφορίες αυτές που δεν ενδιαφέρουν τους περισσότερους καταναλωτές. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πράξη δεν μπορεί να έχει το προφίλ το διατροφικό, ενώ η βιομηχανία είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Και αυτό είναι εις βάρος και της βιομηχανίας και της οικονομίας και των πολιτών. Μπορείτε να μας πείτε στο δικό σας χωρτοφυλάκιο πού θα μειώσετε αυτό το 25% και ποιος θα το ελέγχει και πότε. Και είστε πρόθυμος να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για να δίνετε πληροφορία ε, από εκεί στους καταναλωτές για να μην πλημμυρίζετε τις ετικέτες με αυτές τις πληροφορίες. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο για να ενημερώσουμε τους πελάτες αν έχουμε τη σιγουριά ότι θα φτάσει η πληροφορία σε αυτούς και θα του είναι προσβάσιμη και θα επηρεάσει την απόφασή τους να αγοράσουν. Με αυτήν την αρχή θα κινηθούμε. Προτείνατε παραδείγματο χάρη να πάμε στο ίντερνετ μόνο για τις πληροφορίες. Δυστυχώς διαφωνώ. Γιατί το ίντερνετ, όπως ξέρουμε, δεν είναι προσβάσιμο από όλους πόσοι ξέρουν να πηγαίνουν επιγραμμικά για να βρουν πληροφορίες. Πόσοι γνωρίζουν αγγλικά που είναι και η βασική γλώσσα όπου παρουσιάζονται οι περισσότερες πληροφορίες στο ίντερνετ. Μπορούμε να πούμε ότι ας βάλουμε στο ίντερνετ την πληροφορία και ας την πάρει όποιος θέλει, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο για τον καταναλωτή και βραχικυκλώνει και τις ευθύνες μας έναντι των καταναλωτών. Πρέπει να φροντίσουμε να ενημερωθούν οι καταναλωτές. Αυτό θα φροντίσουμε. Εγώ θέλω ενημέρωση όταν πάω να αγοράσω κάτι. Και μερικές φορές αγοράζω πράγματα κοιτάω ένα προϊόν και κοιτώ και τα συστατικά, την πληροφορία του και μετά αποφασίζω αν θα το αγοράσω ή όχι. Αυτή η προσβασιμότητα θα πρέπει να υπάρχει στους καταναλωτές όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω ένα προϊόν και μετά λέω ας το αφήσω και μετά να πάω σπίτι να κοιτάξω το ίντερνετ, να κοιτάξω την ενημέρωση και να επανέλθω μετά να το αγοράσω. Δεν είναι βολικό αυτό για να σας πω την αλήθεια ούτε καλό για τον καταναλωτή. Πολλέ οι αντιδράσεις, αλλά εγώ νόμιζα ότι ζούσαμε σε ένα σύγχρονο κόσμο και κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Είπατε ότι θέλετε μεγαλύτερη πρόληψη και μεγαλύτερη πληροφόρηση για τα παιδιά. Ωραία είναι αυτά που λέτε. Εγώ εργάζομαι σε ένα Ινστιτούτο ε, εικονική ε, γνώσης και κάνουν και διδακτορικό επιστήμονες για τη γνώση και τις προφορίες σε σχέση με τα τρόφιμα και θέλουμε έτσι να φτιάξουμε κάποια μαθήματα, διδακτέα ύλη για τα δημοτικά σχολεία για τα παιδιά, για να ε, ενημερώνουμε στα σχολεία και να μπορούν τα παιδιά να ε, διαπαιδαγωγούν ξανά από την αρχή τους γονείς τους ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες. Και έτσι και το κόστος ε, αυτό θα μειωθεί. Εσείς θα μας υποστηρίξετε για τη μαγειρική. Τι να σας υποστηρίξω. <laughs> ναι, έλεγα, θα μας υποστηρίξετε. Τέτοια, ένα πανεπιστήμιο παιδικό για μαγειρική. Ε, με ιδέες, όχι με χρήματα. Kitchen University. children. Kids, children, παιδιά, να μαθαίνουν στους γονείς τους να μαγειρεύουν, να μην τρώνε ό,τι να είναι. Children's University of Cooking, Ακαδημία Μαγειρικής για παιδιά. Okay. Um, uh, well, thank you very much. grand idea, I think. Μεγάλη ιδέα. Um, uh, uh, but I, believe, especially in... Πιστεύω και ιδιαίτερα στη χώρα μου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων, ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα, διδάσκουν στα παιδιά να μαγειρεύουν. Πριν καν φτάσουν στο πανεπιστήμιο μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Σας είπα και με αυτό το ερώτημα επανέρχομαι σε αυτά που είπα προηγουμένως ότι θα συνεργαστώ και με την κυρία Βασιλείου θα συνεργαστούμε ώστε η εκπαίδευση και οι γενικότερες δεξιότητες της καθημερινής ζωής να προωθηθούν στα σχολεία μας. Η Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση από την Επιτροπή Γεωργία. Ε, η Ελίζα Γέγκλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιο Επίτροπε, η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών. Πολλά είπατε σχετικά αφενός, αλλά αφετέρου θέλω να ρωτήσω και για τις εισαγωγές. Μας λέτε ότι η προστασία των ζώων θα πρέπει να είναι για όλα τα ζώα. Βεβαίως και θα σας υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι για μας σημαντικό επίσης την κλωνοποίηση των ζώων και εδώ θα ήθελα να προσθέσω και τα διπλώματα εύρηση τεχνίας. Θέλετε να δραστηριοποιηθείτε πολύ νωρίς και για τη στρατηγική της υγείας ε, των ζώων. Ποιοι είναι οι στόχοι σας συγκεκριμένα όμως. Και κύριε υποψήφιε, για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες είστε πρόθυμος να επιβάλλετε τα ειδικά μας υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα και να τα κάνετε και γνώμονα ε, και για ελέγχους και στη συνέχεια για διοδότηση κυκλοφορίας των προϊόντων αφόρων. Ευχαριστώ πολύ. As Σας είπα και προηγουμένως ότι η κλωνοποίηση πρέπει να εξεταστεί ως ξεχωριστό συγκεκριμένο θέμα και να εστιάσουμε την προσοχή μας αυτή ως, όχι ως τμήμα μιας άλλης οδηγίας όπου αναφέρεται σε μερικές παραγράφους. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρω ότι και αφού το έχω συζητήσει και με τις υπηρεσίες μου βεβαίω. δεν τα εφευρίσκω όλα αυτά ότι μέσα σε ένα χρόνο θα σας υποβάλουμε έκθεση για το θέμα της κλωνοποίησης και μετά όλοι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και τις επιπτώσεις του τομέα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω την έκθεση της Επιτροπής Διοντολογίας, γνωρίζω ότι ακόμα και η ίδια η ΕΦΣΑ λέει ότι ναι μεν τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα είναι ασφαλή αλλά η ίδια η ΕΦΣΑ αναγνωρίζει ότι το θέμα είναι προβληματικό της εξαιτίας ακριβώς της κλωνοποίησης και η προστασία των ζώων είναι και αυτή τμήμα των αρμοδιοτήτων μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό από κοινού να εξετάσουμε το θέμα για να καταλήξουμε στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από την Επιτροπή Γεωργίας. Κυρία ε, ε, Γαρσία Πέρες, ευχαριστώ. Για την ε, υγεία των ζώων και την προστασία των φυτών, τα μεταλλαγμένα κτλ. γίνεται λόγος για κάποιες προδιαγραφές πολύ υψηλότερες σε μερικές περιπτώσεις από τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και αυτά που χρησιμοποιούν περισσότεροι ανταγωνιστέ μα. Η κατάσταση αυτή έχει αρνητικέ συνέπειε στην ανταγωνιστικότητα τη γεωρική μα παραγωγή. Δέχομαι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε του κανόνε παιχνιδιού των διεθνών οργανισμών για το διεθνέ εμπόριο. Αλλά ποια μέτρα θα πρέπει, σκέφτεστε να λάβετε στα πλαίσια αυτά για να μην συνεχίζουν να χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους οι Ευρωπαίοι γεωργοί. Αριστερά σας ήταν ο μιλήτρια. Κοιτάξτε και λιγάκι προς τα αριστερά, μπορεί και να τη βλέπατε. I don't believe that our standards should be those... Δεν πιστεύω ότι τα πρότυπα μας είναι, είναι χειρότερα από των ανταγωνιστών. Θεωρούμε ότι τα πρότυπα μας πρέπει να βασιστούν στα... σε επιστημονικές γνώσεις, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι μετά οι ανταγωνιστές μας δεν θα έχουν πλεονέκτημα στην αγορά μας. Δεν θα μπορούν να εξάγουν με χαμηλότερα πρότυπα μετά στην αγορά μας. Αυτό πρέπει να διατηρήσουμε ως αρχή, ότι οτιδήποτε εισάγεται θα πρέπει να σέβεται τα ίδια πρότυπα με οτιδήποτε παράγεται στην Ευρώπη και μετά τα πρότυπα πρέπει να είναι τα δικά μας πρότυπα με βάση τα όσα μας λένε οι επιστημονικές σύμβουλες για τα επίπεδα ασφάλειας των καταναλωτών μας. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ερχόμαστε στον τέταρτο γύρο ερωτήσεων. Πρώτος ο Λαφ Μικολάσικ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την... τις ξεκάθαρες απαντήσεις που μας δώσατε μέχρι τώρα ως κύριος εισηγητή για την οδηγία της Κομισιόν και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για, τις, για ανθρώπινα όργανα για μεταμοσχεύσεις. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμφωνία και στην πρώτη ανάγνωση υπό Ισπανικής Προεδρίας. Αυτό το χρειάζεται η Ευρώπη. Εγώ και οι σκιώδεις συνεισηγητές είμαστε υπέρ της αρχής του άρθρου 13 για εθελοντική και μη αμοιβόμενη δωρεά. Για να μην έχουμε εμπόριο ή εμπορική συναλλαγή των οργάνων και για να σεβαστούμε και την ακαιρεότητα του ασθενούς, θέλω να σας ρωτήσω αν είστε διατεθειμένος να υποστηρίξετε αυτή την αρχή της μη αμοιβόμενης και εθελοντικής δωρεάς και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Απάντηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα με την αρχή αυτή και μπορώ να σας πω ότι υποστηρίζω πλήρως την εθελοντική και μία αμοιβόμενη δωρεά. Σας ευχαριστώ για την ξεκάθαρη απάντησή σας. Για να εξασφαλιστεί μια ενιαία προσέγγιση σε όλους τους τομείς της υγείας. Το ερώτημα είναι το εάν θα θέλατε να εφαρμόσετε αυτή την αρχή και σε άλλες οδηγίες που ήδη υφίστανται, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα, για την οδηγία για ιστούς και κύτταρα του 2004. Είστε διατεθειμένος να επανέλθετε. Απάντηση. Να σας το πω ως εξής. Θα είμαι ιδιαίτερα ανοιχτό για οποιαδήποτε συστάσεις υπάρξουν από εμπειρογνώμονες όπως εσείς για να εξασφαλίσω ότι οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να εδρεωθεί αυτού του είδους η αρχή εντός όλων όσων κάνουμε και να είμαστε συνεπείς, γιατί και η συνέπεια είναι βασικό τμήμα της πολιτικής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε συνεπείς σε όλες τις αρχές που ανακοινώνουμε. Θα βασιστώ στις συμβουλές σας. Ευχαριστώ πολύ. Από τους μη εγγεγραμμένους δεν είχαμε καμία δήλωση ονόματος. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χόρστ Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντάλι, θα ήθελα να εκφράσω εδώ την ικανοποίησή μου για τα όσα μας είπατε για τα κλωνοποιημένα ζώα. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω σοβαρά να εξετάσετε και να φροντίσετε αυτά που θα φέρετε εδώ να εξετάσουμε εμείς να μην είναι έκθεση αλλά είναι πρόταση για πολιτική. Τώρα θα έχουμε και πολλές ε, νέες ρυθμίσεις μετά από μεταβατικές περιόδους και πολλές διατάξεις καταφέραμε να προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται ορισμένες ε, ε, παρατάσεις μέχρι το 2013 ε, λέτε οι μεταβατικές περίοδοι. Εγώ δεν το θεωρώ σκόπιμο κάτι τέτοιο. Εσείς είστε πρόθυμος. Τώρα, ε, μετά τις προθεσμίες με το 2013 θέλετε μαζί με το Κοινοβούλιο να ελέγξουμε αν χρειάζεται αλλαγή ο κανονισμός, τροποποίηση. Δεύτερη ερώτηση. Εδώ και χρόνια γονιζόμαστε για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Όλο νέα ντοσιά έχουμε νέου φακέλου. Πώ θα καταπολεμήσουμε τι ελλείψει κτηνιατρικών φαρμάκων. Έχετε καμιά πρόταση επιτέλου να λύσουμε αυτό το θέμα. What we will be doing on an... Το τι θα κάνουμε ε, για την κλωνοποίηση, είπα και πριν ότι θα ρίξουμε φως στο θέμα θα το φωτίσουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ελπίζω, βέβαια και οριζοντίως με άλλες γενικές διευθύνσεις και άλλους επιτρόπους για να ε, υποβάλουμε εν τέλει μια συνολική πρόταση και να καταθέσουμε εν πάση περιπτώσει μια πρόταση που να συζητηθεί. Και πάλι λέω ότι δεν πιστεύω ότι θα παίρνουμε αποφάσεις πριν να έλθουμε σε εσά για να τα συζητήσουμε μαζί σας. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να τηρήσω πάντοτε την αρχή, να βάζω το κοινοβούλιο στην διαδικασία λήψης απόφασης όσο γίνεται νωρίτερα. Προτιμώ δηλαδή να διαθέσω χρόνο να συζητήσω μαζί σας από πριν παρά να χάσω χρόνο αντιμαχόμενο σε εσά αργότερα, επειδή μπορεί να μην σα αρέσει η πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν και το επίπεδο και η ουσία του εγγράφου θα πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να συζητηθεί με καρποφόρο τρόπο και θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι στις διάφορες θέσεις που θα λάβουμε όλοι δηλαδή οι συνομιλούντες γύρω από το τραπέζι και πολύ καλύτερα θα μπορούμε να καταλήγουμε σε μια συμφωνία. Για τα κτηνιατρικά φάρμακα, εγώ θα πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν έχω πολύ χρόνο για να σας πω τώρα. Είπα ποια, ποιες είναι οι αντιστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό που χρειάζεται είναι να φροντίσουμε ώστε όλα τα σχετικά να είναι καλά μελετημένα και να μπορέσουν να επιβληθούν σωστά. Ο κ. Σνέλχαρτ, ευχαριστώ κύριε Νταλή. Έρχομαι στην δεύτερη ερώτησή μου για τους σχετικούς κανονισμούς, τους οποίους έχουμε παρατείνει μέχρι το 2013, που νομίζω όμως ότι δεν αποτελεί λύση. Παρακαλώ να εξετάσετε σε συνεργασία με την Ευρωβουλή να γίνονται κάποιες αλλαγές έστω καλοπιστικέ των κανονισμών, κάτι το οποίο έχει αρνηθεί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε εσεί. Μιλάτε για τις ε, δοκιμές, για τα πειράματα επιζών. Μιλώ για τον κανονισμό περί υγιεινής, κανονισμό περί που χρονολογείται το 2006. θα χρειαστεί να το μελετήσω βαθύτερα πριν να μπορέσω να σας δώσω μια ουσιαστική απάντηση. Όπως έδωσα σε προηγούμενες απαντήσεις. Η κυρία Για την πολιτική τροφίμων. Στόχος της Ευρωπαϊκής ε, Πολιτικής Προστασίας Καταναλωτών είναι ο καταναλωτής να είναι ελεύθερος να επιλέγει. Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί θέμα με κάποιες απομιμήσεις τροφίμων με ε, μορφή τυριών ή με μορφή ε, ε, χειρομεριού λοιπά, τα οποία παριστάνουν κάτι που δεν είναι. Παραπλανούν λοιπόν τους καταναλωτές. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς περιέχεται μέσα στο τρόφιμο το οποίο καταναλών. Θα μας υποστηρίξετε στην πρωτοβουλία για την προστασία των καταναλωτών απέναντι σε τέτοιες απομιμήσεις ε, τροφίμων. Η θέση μου για τα προϊόντα τέτοια απομίμησης είναι ότι αποτελούν απάτη. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από τα χέρια μας για να φροντίσουμε να μην εξαπατώνται οι καταναλωτέ μας. Να μην θεωρούν ότι αγοράζουν κάτι όταν αγοράζουν κάτι άλλο. Να μην αγοράζουν κάτι που θεωρούν ότι είναι καλό για την κατανάλωσή του, όταν στην πραγματικότητα μπορεί να τους σκοτώσει. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι όντω θα κινηθώ και θα κινηθώ ταχύτατα για να διασφαλίσω ότι θα υπάρξει επαρκή σήμανση των προϊόντων αυτών στον τομέα. Σας ευχαριστώ για την ξεκάθαρη απάντηση και δήλωση. Εν προκειμένου έχω και μια ερώτηση πάντοτε για τον ελεύθερο καταναλωτή. Μιλήσαμε για την ενημέρωση. Η ερώτησή μου είναι θα υποστηρίξετε την πρόταση να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ή και εθνικές ιστοσελίδες του διαδικτύου δηλαδή που να ενημερώνουν ουδέτερα σχετικά με διάφορες θεραπείες νόσων ή ασθενειών, επιπροσθέτως εκείνων των ιστοσελίδων που ε, δίνονται από διάφορους ε, παρασκευαστές φαρμάκων. Κυρία Βασκέρμπερ, γνωρίζετε ότι, το, τον κανόνα ότι η συμπληρωματική ερώτηση πρέπει να αναφέρεται στην πρώτη ερώτηση. Η δική σας ήταν τελείως διαφορετική. Δεν χρειάζεται να απαντηθεί λοιπόν και προχωρώ αμέσως στην κυρία Σαλντεμόζ. Øh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ σε αυτό που είπατε, ότι θέλετε να υπερασπίζεστε σωστά τον καταναλωτή. Τι σημαίνει αυτό. Μπορείτε να δεσμευθείτε, να υποσχεθείτε ότι όταν καταθέτετε πρόταση για τους καταναλωτές δεν θα ξεχάσετε κανένα Ευρωπαίο καταναλωτή, δεν θα αφήσετε στην άκρη κανένα καταναλωτή και θα λαμβάνετε τους πάντες υπόψη όταν κάνετε συστάσεις για εναρμονίσεις για προϊόντα καταναλωτικά. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι θέλετε ελάχιστη εναρμόνιση ή σε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Μήπως χρειάζεται όμως η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών of Για την οδηγία των δικαιωμάτων καταναλωτών. Νομίζω ότι αυτή έχει περάσει στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Ρέντινγκ τώρα. Σε ό,τι αφορά πάντως το θέμα της εναρμόνισης, είτε ελάχιστης είτε πλήρους, που ε, πιστεύω ότι συζητείται εντατικά τώρα, η γνώμη μου είναι μάλλον ότι πρέπει κανείς να προχωρήσει προσεκτικά η εναρμόνιση, όπως είπα και πριν. η συνοχή είναι το κλειδί. Δεν μπορούμε να λέμε ένα πράγμα σε ένα τομέα και κάτι διαφορετικό σε άλλο τομέα. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί, συνεπείς στις σκέψεις μας. Εάν πιστεύουμε στην ενιαία αγορά, και πιστεύουμε ότι ορισμένες απαιτήσει, κυρίως ό,τι αφορά δικαιώματα των καταναλωτών, είναι σημαντικές για την ενιαία αγορά, τότε πρέπει να κινηθούμε με τρόπο που θα εναρμονίσει την ενιαία αγορά όσο αυτό είναι δυνατό. Όπως είπα, το θέμα των προδιαγραφών για μένα είναι, δεν είναι θέμα διαπραγματεύσεων τι μπορώ να δώσω και τι μπορώ να πάρω. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το σωστό επίπεδο προδιαγραφών που αναμένει ο Ευρωπαίος καταναλωτής είτε βρίσκεται στην Φιλανδία είτε στη Βουλγαρία. Ποιο είναι το επίπεδο προδιαγραφών που πρέπει να προσφέρουμε στον καταναλωτή μας. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επιδεκτικοί σε αυτή την έννοια. Όταν μιλεί κανείς για κεκτημένα δικαιώματα και νομίζω ότι οι οργανώσεις των καταναλωτών τώρα έχουν πάρει τα όπλα για τα θέματα αυτά. Η κτήση δικαιωμάτων είναι βεβαίως δημοκρατική διαδικασία. Υπάρχουν όμως και πολλά ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από την έννοια αγορά. Και χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια εξισορρόπηση των ενδιαφερόντων αυτών. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τεθεί επιτάπητο. Τα ωφέλη τη ενιαία αγορά, Υπάρχουν ωφέλη την ενιαία αγορά ή όχι. Ναι, ευχαριστώ. Αλλά ε, δεν νομίζω να έχω περισσότερη πληροφόρηση. Δεν πρόκειται για την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Εγώ σας μίλησα για τις μελλοντικέ προτάσεις νομοθεσίας που θα κάνετε για την προστασία των καταναλωτών. Τι προτάσεις θα κάνετε προς πλήρη εναρμόνιση ή προς την ελάχιστη εναρμόνιση. Αντιλαμβάνομαι την απάντησή σας ως εξής όμως, ότι θα υπάρχουν καταναλωτές Ευρωπαίοι που δυστυχώς δεν θα μπορούν να υποφελούνται από δικαιώματα που ήδη θα θεωρούν και εκτιμένα στις χώρες τους. Απάντηση. Εάν κληθώ να λάβω αποφάσεις για νομοθεσία που πρόκειται να επηρεάσει την ενιαία αγορά και επιθεμάτων που θα είναι σημαντικά για την αγορά των καταναλωτών. Θα προτιμήσω να ωφελήσω την ενιαία αγορά, διότι πιστεύω ότι εν τέλει από αυτό θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Εάν αυτό σημαίνει, σημαίνει μάλλον εναρμόνιση, τότε θα αποφασίσω υπέρ της εναρμόνισης. Και νομίζω ότι εκεί εντοπίζονται και τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι πολιτικοί. Μιλούμε για μια και για, κοινότητες με ποικίλε παραδόσεις που έχουν διαμορφωθεί μέσα στο χρόνο και θα έχουμε περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να συμβιβαστούμε έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια κατάσταση που να ωφελήσει όλους και να του ωφελήσει πραγματικά. Εάν πιστεύω ότι η αγορά είναι εποφελής, μπορεί κανείς να χάσει κάποια δικαιώματα, από την, άλλη, από την άλλη μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι προσιτά και σε τιμές ε, που καθιστούν προσιτά τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν θα είναι ή το ένα ή το άλλο. Νίκολσον. Η Ευρώπη εισάγει σημαντικές ποσότητες προϊόντων από όλο τον κόσμο. Τα ε, προϊόντα των Ευρωπαίων ε, γεωργών, αγροτών, παραγωγών σέβονται αυστηρές προδιαγραφές. Τι θα κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από άλλες χώρες να υπακούν στις ίδιες προδιαγραφές θα υπερασπιστείτε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στον ΠΟΕ και τι θα κάνετε για τις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή οργανισμών στην Ένωση. Για παράδειγμα, βόλιο κρέας από την Βραζιλία, που δεν ε, ανταποκρίνεται στις αυστηρές προδιαγραφές τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και τι θα κάνετε και με την ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων που μέχρι τώρα δεν έχει εξυπηρετήσει. Όλα αυτά σε δύο λεπτά. <laughs> Για να απαντήσω. Κοιτάξτε, επαναλάβω κάτι που είπα. Η βασική αρχή είναι ότι το τρόφιμο που θα εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι βραζιλιάνικο βόλιο κρέας, θα πρέπει να έρεται στο επίπεδο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ε, δεν έχω αναλάβει ακόμα το αξίωμα, αλλά πάντως εάν το αναλάβω δεν θα δεχτώ ή οδήποτε τρόφιμο ή ασδήποτε μορφής που να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι υποδέστερης ποιότητας ή εν πάση να μην συμμορφώνεται με τις ποιοτικέ προδιαγραφές που οφείλουν να σέβονται τη δική μας παραγωγή. Αυτή είναι η βασική αρχή. Γνωρίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι, για παράδειγμα όταν μιλάτε για το βόλιο κρέας από τη Βραζιλία, είναι γεγονός ότι το FIO e ο οργανισμός των ε, κτηνιάτρων, έχει επιβεβαιώσει τον τόπο προέλευσης, Βραζιλία. Εφόσον το προϊόν αυτό έχει πιστοποιηθεί στη Βραζιλία ως ανταποκρινόμενος προδιαγραφές μας, τότε μπορεί να μπει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για την σήμανση των προβάτων. Όπως ξέρετε, έχει αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα από την πρώτη του μηνός. έχει εφαρμοστεί και για κάποιο διάστημα σε πολλές άλλες χώρες. Άλλες χώρες καθυστερούν ακόμα. Όπαντος η οδηγία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Εάν δούμε ότι κάποια πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες συνέπειες. Αλλά για την ώρα η θέση είναι ότι εφαρμόζεται η οδηγία επισήμανση των προβάτων και αυτή είναι η πολιτική την οποία ασκούμε. Μάρτιν Χόισλινγκ. Ο κύριος Μπαρόσο πρότεινε να αναλάβουν οι ίδιες τις αποφάσεις, οι χώρες μέλη να αναλάβουν τις ε, αποφάσεις, να αναλάβουν τις αποφάσεις σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ε, πώς το βλέπετε αυτό. Είναι δύσκολο βέβαια μέσα στο μικρό περιορισμένο σχετικά γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης να μπουν σύνορα στην ενδεχόμενη μόλυνση των εισαγωγικών ε, του γενετικού υλικού από τέτοια προϊόντα. Δεύτερο, το Κοινοβούλιο συμφωνεί σε ό,τι αφορά την προστασία των σπόρων. Δέχεστε την ε, θέση του Κοινοβουλίου εν προκειμένου και θα κάνετε πάντο δυνατόν ειδικά για ε, το υλικό σποράς ε, να έχουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη μόλυνση από γενετικά τροποποιημένα υλικά. Πάλι για το ίδιο θέμα από τις λίγες εβδομάδες που έχω ε, αρχίσει να ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, ακούω πολλές απόψεις που δεν είναι ομοιομορφές, δεν είναι όλες εν, ενιαίες, ε, αποκλίνουν και μέσα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται να συζητηθεί επαρκώς θα το συζητήσετε κι εσείς, τα γάματα φόμικρον και εμείς το ίδιο. Και θα συζητήσω κι εγώ μαζί σας τα θέματα που σχετίζονται με τους γεννητικά τροποποιημένους οργανισμούς και ελπίζω ότι εν τέλει θα μπορέσουμε να λάβουμε ταχαίως αποφάσεις. Είπα και πριν ότι αυτό το επίπεδο αβεβαιότητας που ε, υπάρχει για ε, τα ζητήματα αυτά δεν ωφελεί κανένα. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε όντως με κάποια ταχύτητα για τα θέματα αυτά, να εξετάσουμε ε, ε, ενδεχόμενες λύσεις που να είναι και ρεαλιστικές αλλά και ασφαλείς, γιατί η ασφάλεια είναι εκείνη που πρωτίστως ενδιαφέρει και που ο καθένας να μπορεί να δεχτεί ότι είναι ο σωστός τρόπος Πέμπτος γύρος ερωτήσεων. Φιέλνερ. σε ευχαριστώ. Κύριε Ντάλη, χαίρομαι που θέλετε να δώσετε εξουσία στους καταναλωτές μέσω ενημέρωσης και επιλογής. Το ίδιο ελπίζω να κάνετε και με τους ασθενείς. Και να είστε προετοιμασμένος να έχετε πολλούς νέους εχθρούς από τα κράτη-μέλη πάντως. Πρέπει να είστε σκληρός πάντως προς όφελος των ασθενών που έχουν ιδιαίτερα χρόνιες ή σπάνιες ασθένειες και οι νέες θεραπείες είναι ζήτημα θανάτους. Γι' αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο για 8 χρόνια προτείνουμε αυτή την πρόταση. Θέλετε εσείς να επανεξετάσετε αυτό το πακέτο. Τι σημαίνει επανεξέταση και τι ελπίζετε μετά από αυτή την επανεξέταση. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας πάντως ότι τα λεγότερα αμφιλεγόμενα τμήματα του πακέτου δεν θα πρέπει να περιμένουν τα περισσότερα αμφιλεγόμενα για να περάσει το πακέτο. Αλλά η ενημέρωση του ασθενούς δεν θα πρέπει να θυσιαστεί και να καθυστερήσει πέραν του απαραίτητου. for Βρίσκομαι στην πολιτική ζωή για πολλά χρόνια και πάντα ήμουν σε θέσεις όπου χρειάστηκε ο ίδιος να υιοθετήσω πολύ δύσκολες θέσεις στη χώρα μου περνώντας φορολόγηση ως υπουργό Οικονομικός στην Μάλτα απελευθέρωση της οικονομίας όταν ήμουν υπουργό Οικονομικών και Εμπορίου και απελευθερώντας πολλούς άλλους τομείς στην Μάλτα. Δυστυχώς σε τέτοιες θέσεις το να κάνει κανένας εχθρούς είναι τμήμα της δουλειάς του. Δεν με φοβίζει λοιπόν αυτό ούτε θα με αποσταθεροποιήσει από τα όσα εγώ πιστεύω πρέπει να γίνουν για τους καταναλωτές. Στον κόσμο αυτό κάνει κανένας πολλούς εχθρούς για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Εάν ξέρετε όμως ότι η κατεύθυνσή σας είναι η σωστή, τότε πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει κανείς. Για το αποτέλεσμα της επανεξέτασης του, των προτάσεων για ενημέρωση των ασθενείων. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να αναμένω την επανεξέταση. Για πάλι, αυτό παρακαλώ υπομονή. Συμπληρωματικό ερώτημα. Είμαι υπομονετικός, αλλά γιατί χρειάζεται επανεξέταση. Αυτό μπορείτε να το σχολιάσετε, γιατί ελπίζουμε έτσι να κατανοήσουμε και το σκεπτικό σας. Και χαίρομαι που έχουμε ένα υποψήφιο επίτροπο που είναι έτοιμος να περάσει στη μάχη, γιατί αυτό χρειάζεται. Και Θέλουμε ένα αποτέλεσμα στον τομέα αυτών που να μην είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής, γιατί συχνά αυτό συμβαίνει σε πολύ αμφιλεγόμενα θέματα. Ελπίζω πάντως να δώσετε μάχη, αλλά πέστε μας γιατί χρειάζεται επανεξέταση. Σε αυτή την επανεξέταση θα εξασφαλίσουμε ότι ίσως υπάρξει μεγαλύτερη διασάφηση του τι είναι ενημέρωση και τι είναι διαφήμιση. Αυτό είναι σημαντικό για να μην διατρέξουμε τον κίνδυνο. Κόσμος κάποια στιγμή στη ζωή τους που είναι ευάλωτοι γιατί υποφέρουν από μία ασθένεια να υποχρεωθούν να αγοράσουν προϊόντα που τελικά ίσως δεν είναι καλά για αυτούς. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Θα επιμείνω λοιπόν ώστε να υπάρξει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση και στη διαφήμιση. Και μετά πρέπει να εξασφαλίσουμε ποια είναι η πληροφορία που χρειάζεται ο ασθενής, ποια είναι η προοπτική του ασθενούς, πότε χρειάζεται την ενημέρωση. Εγώ προσωπικά φοβάμαι μήπως βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις για την υγεία τους χωρίς τη συμβουλή των επαγγελματιών του κλάδου. Αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό πρέπει να το συζητήσω μαζί σας για να δούμε ποια θα είναι η διαχωριστική γραμμή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ευθύνη της κυρία, Στρέλα είναι γνωστές οι ευθύνες της ε- ε- Ευρώπης και η συνθήκη της Λισαβόνας εισαγάγει δυνατότητα ανάληψη δράσης για συγκεκραμένες ασθένειες. Σε ποιες ασθένειες θα επικεντρώσετε την προσοχή σας και θα ήθελα να αναφερθείτε στο εάν οι ρευματοπάθειες θα είναι τμήμα αυτής της προσοχής. The now. Η άποψη που, στην οποία κατέληξα μέχρι τώρα είναι ότι θα επικεντρωθώ κυρίως όχι σε συγκεκριμένες ασθένειες, αλλά σε ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας. Με περιορισμένους πόρους που έχουμε, θεωρώ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πηγές ασθενειών που αφορούν πολλές ασθένειες. Δεν είμαι ιατρός, αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι που επηρεάζουν πολλές ασθένειες. Παχυσαρκία παραδείγματος χάρη που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο, μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοαγγειακά και ασθένειες. Δηλαδή να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες ασθένειες, τι να σας πω θεωρώ ότι θα μας δώσει μόνο αυτό μία βραχυπρόθεσμη λύση. Ενώ αν επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε γενικότερους παράγοντες που επηρεάζουν πολλές ασθένειες θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και η προσπάθεια στην, για την πρόληψη θα μας οδηγήσει σε πιο καλύτερα αποτελέσματα. Και έτσι θα έχουμε πιο εύκολα αποτελέσματα αν το συγκρίνουμε αυτό με συγκεκριμένη περίθαλψη ή θεραπεία και θεωρούμε ότι σε αυτούς τους τομείς εμείς Κομισιόν και εσείς Κοινοβούλιο μπορούμε από κοινού να κάνουμε προσπάθεια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης για να καταπολεμήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν την γενικότερη υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα και αν έχουμε προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου και άλλες μεμονωμένες ασθένειες. Ε, ήταν ευρύτερη ερώτηση, αλλά θα το ξαναδούμε αυτό αργότερα. Ε, κυρία Ρούλε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντάλη, ε, τονίζετε την επιβολή του νόμου και τον ενημερωμένο ε, καταναλωτή. Ωραία είναι αυτά, αλλά πώς ελέγχετε η αγορά, πώς παρακολουθείτε. Γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν πράττουν αυτά που έχουν δηλώσει ως καλές προθέσεις. Τι θα κάνετε, ας πούμε, ε, και το είδαμε αυτό και στα άλλα αγαθά, ε, ε, στα βιομηχανικά αγαθά και όταν έχουμε προβλήματα με ελαττωματικά παιχνίδια ή ελαττωματικά άλλα βιομηχανικά προϊόντα, τι κάνετε. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πάρα πολύ κρυφό ποιοι συνεδριάζουν εκεί, ποιοι συμμετέχουν και ποιοι αποφασίζουν. Τι θα κάνετε για να είναι πιο δημόσια τα πράγματα εκεί και τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται. Και επίσης υπάρχουν διάφορες επιτροπές Πιστοποίηση, και για αυτές γνωρίζει πάρα πολύ λίγα το Κοινοβούλιο. Και πάλι εκεί δεν είναι ισορροπημένη η σύνθεση. Για παράδειγμα, είναι πολύ λίγοι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πάρα πολύ λίγε οργανώσει καταναλωτών. Τι θα κάνετε εσεί προ την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε και σε αυτούς τους ε, ε, φορείς πιστοποίηση να είναι καλύτερη και πιο ισόρροπη η εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων. θα εξετάσω όλα αυτά τα θέματα για να εξασφαλίσω ότι οτιδήποτε τελικά θεσπίσουμε ως μηχανισμούς για να μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε θα λειτουργήσουν σωστά. Σε τι αναφέρατε, αν υπάρχει μεροληπτική θέση θα πρέπει να βρούμε ποια είναι και να τη διορθώσουμε γιατί χρειάζεται αντικειμενική θέση και συμβουλή το ίδιο ισχύει και για τη διαφάνεια. Πιστεύω ότι αυτή η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σέβεται τη διαφάνεια την οποία πρέπει να εφαρμόσει συνεπώς σε οτιδήποτε κάνουμε. Βεβαίως και εδώ με κάποιες επιφυλάξεις, διότι δεν μπορείτε να είστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου θα πρέπει να σεβαστείμε κάποιου είδους εμπιστευτικότητα στην διαδικασία στην οποία έχουμε. Για την εποπτεία. Πρόκειται για ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών και εξασφάλιση ότι οι δυνατότητες των κρατών μελών σέβονται το επίπεδο που απαιτείται και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ανθρωπίνων πόρων και την μηχανική και τεχνολογική δυνατότητα που υπάρχει, καθώς επίσης και στο επίπεδο των ανθρωπίνων πόρων που είναι σε ενέργεια στον τομέα. Και εμείς ως Κομισιόν δεν θέλουμε να αναλάβουμε την εποπτεία, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη η δυνατότητα που έχουν είναι στα σωστά επίπεδα. Ε, Πάλι για, τους, για τις επιτροπές τυποποίησης. Έχουμε πολλά, πολλές οδηγίες, οδηγίες που βασίζονται σε αυτή τη new approach και η τελευταία οδηγία ήταν για τα παιχνίδια. Το πρόβλημα είναι όταν έχουν εγκριθεί και ψηφιστεί αυτές οι οδηγίες δεν μαθαίνει το κοινοβούλιο τι γίνεται. Για παράδειγμα, για τον θόρυβο δεν έχουμε τιμές κατόφλια για ε, την ε, για τον θόρυβο, Επίση για διάφορε αρωματικές ουσίε. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσετε αν αυτή η προσέγγιση είναι σωστή και πώς μπορεί να αποκατασταθεί η διαφάνεια και πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να ενισχυθεί και να μην αποδυναμωθεί η θέση του με αυτή την new approach, την νέα προσέγγιση. Απάντηση. Όταν λαμβάνεται μια αναλαμβάνεται μια δράση, όπως για τα παιχνίδια. Συνήθως μετά ακολουθεί η θέσπιση προδιαγραφών. Και ζητούμε από την ΕΦΣΑ να θεσπίσει προδιαγραφές. Και τώρα θα κάνω λίγη αυτοδιαφήμιση, δηλαδή για διαφήμιση για, για αυτά που χρειάζομαι. Θα ζητήσουμε από την ΕΦΣΑ, χρειαζόμαστε μόνο και περισσότερη χρηματοδότηση. Γιατί χρειαζόμαστε ταχύτητα αποφάσεων και ακρίβεια αποφάσεων και με το πιο ανεξάρτητο τρόπο. Αλλά ας βάλουμε και το χέρι στην τσέπη και ας χρηματοδοτήσουμε με το σωστό τρόπο τις οργανώσεις αυτές ώστε ε, να μπορέσουν πραγματικά να αποδώσουν σε αυτά που τους ζητούμε. Μακλάρκιν. για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Όταν θα περάσει η πρόταση αυτή, οι καταναλωτές θα βρίσκουν πάνω στις ετικέτες των τροφίμων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να κάνουν την επιλογή τους όντας ενήμεροι. Και η συγκήτρια Ζόμερ έχει δίκιο που λέει και για το άρθρο 4 της ε, οδηγίας, του κανονισμού μάλλον, για τα ε, claims, για τους ισχυρισμούς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πώς εσείς θα βρείτε μια ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς με την πληροφόρηση των πολιτών, των καταναλωτών όπως αυτή πρέπει να γίνεται και την ελευθερία επιλογής. Σε όλες τις πρωτοβουλίες είναι η απάντηση που αναλαμβάνουμε για την επισήμανση. Δεν νομίζω ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγόρευσε την διάθεση στην αγορά κάποιες, κάποιου τροφίμου. Σε ό,τι αφορά την επιλογή, λοιπόν, η επιλογή υπάρχει. Εκεί που επιμένουμε είναι αν έχουν επιλογή οι καταναλωτές. Το πρόβλημα δηλαδή είναι εάν αναζητούν πληροφορίες και δεν τις βρίσκουν. Και το καθήκον μας είναι να παρακινήσουμε τους καταναλωτές μας, να τους κάνουμε λόμπι δηλαδή, για να αναζητήσουν τις πληροφορίες αυτές. Αυτή τη στιγμή θα θέλουν τις πληροφορίες, πρέπει να εξετάσουμε αν θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες. Τώρα, είναι πολύ πυκνογραμμένη η ε, πληροφορία και ε, δεν μπορεί κανείς να τη διαβάσει, να την αποκρυπτογραφήσει. Αυτό έλεγα πριν, όταν έλεγα ότι πρέπει κανείς να έχει μια ευγεία σε αυτά τα πράγματα. δεν θα σταματήσουμε καν εκεί, εάν είναι επαρκής η πληροφορία. Αλλά έχουν και την ικανότητα, είναι δηλαδή εκπαιδευμένοι οι πολίτε ώστε να μπορούν να διαβάσουν σωστά τι πληροφορίε αυτέ. Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Και εκεί θα πρέπει να συνεργαστούμε με του καταναλωτέ για να διασφαλίσουμε ώστε οι πληροφορίε που βάζουμε πάνω στα πακέτα είναι, γίνονται και κατανοητέ, Ότι καταλαβαίνουν οι πολίτε, δηλαδή τι διαβάζουν. Smart labeling δηλαδή αλλά και ευανάγνωστες και βέβαια και ένα πρόγραμμα κατάρτισης των πολιτών, των καταναλωτών, ώστε να μπορούν πράγματι να επωφεληθούν από τις προφορίες που λαμβάνουν. Για το ενόπνευμα τώρα, συμπληρωματική ερώτηση, για το 2012 και για την κατάχρηση του ενοπνεύματος χρήση όλων των δυνατών μηχανισμών με εκστατείες ενημέρωσης των πληροφοριών που είναι πολύ καλύτερο παρά με υπερβολική νομοθετική ε, ρύθμιση. Πώς θα ασχοληθείτε με θέματα που έχουν σχέση με το ενόπλωμα στη διάρκεια της θητείας σας. Απάντηση. Εγώ να σας τα πω και με εμπειρία από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν υπουργό υγεία στην Μάλτα και είχα την ειδική αυτή ευθύνη. Η κατάχρηση πνεύματος πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως με μια μεγάλη ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης. Αλλά χρειάζεται και κάποιοι έλεγχοι στην ε, κατάχρηση του αλκοόλ. Για παράδειγμα, ε, μέθη στο τιμόνι. Αυτό βέβαια δεν ανήκει στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Αλλά για να το πετύχουμε πρέπει να αρχίσουμε να σπρώχνουμε όλο και περισσότερο. Δεν θα πούμε στους ανθρώπους να μην πίνουν, αλλά μην κάνουν κατάχρηση. Να μην κάνουν κατάχρηση. Αυτά δεν λύνονται απλώς με ετικετοθεσία στα προϊόντα αναπνεύματο. Πρέπει να είναι ευρύτερα και χρειάζεται να συμβάλλουμε και με κάποιες ανανεωτικές ιδέες. Ευχαριστώ. Ίσια ίσια μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει συμπληρωματική την ερώτησή σας κυρία Μακλάρκιν η ε, κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Ντάλη, εσείς αναλάβατε εκείνο το χαρτοφυλάκιο το οποίο ε, έχει την αμεσότερη σχέση με την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ ε, σοβαρό και οξύνεται. Είναι η αντοχή στα αντιβιωτικά. Όλο και περισσότερα ε, ιδιαίτερα επικίνδυνα μικρόβια σήμερα αντιστούνται σε όλα τα υπάρχοντα αντιβιωτικά. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα γίνεται λόγος για διάφορα φάρμακα, γίνονται διάφορες μελέτες, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν γνωρίζουμε τι αντιβιωτικά συνταγογραφούνται. Ποιος δίνει τι σε αντιβιωτικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα στοιχεία υπόψη μας. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Όταν τα ζώα έχουν καλύτερη υγεία, τότε θα έχουν και οι καταναλωτέ καλύτερη υγεία καταναλώνοντας το κρέας τους. totally agree, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω, το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι χρειαζόμαστε πιο υγιή ζώα για να μας δίνουν πιο υγιεινά τρόφιμα. Όντω, θα εργαστώ προ την κατεύθυνση αυτή και αυτό άλλωστε ε, συνεχίζει την παράδοση του παρελθόντο. Οι υπηρεσίε μας έχουν εργαστεί με τρόπο πάρα πολύ σκληρό ε, ως τώρα για να ε, θέσουν τι κατάλληλε προδιαγραφές και πρότυπα στα κατάλοιπα φαρμάκων στα προϊόντα ζωικής πρόέλευση για τους ελέγχου που γίνονται λοιπόν και την ανείχνευση τέτοιων καταλήπων. Αυτό είναι ένα τομέα όπου πραγματικά εργαζόμαστε ε, και πρέπει να προχωρήσουμε. Ερχόμενος τώρα στη συνταγογράφηση των αντιβιωτικών και πόσα αντιβιωτικά γράφονται κτλ. Και πάλι εδώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να το κοιτάξουμε και επίσης πώς θα συντονίσουμε ε, τη δράση μας με την Επιτροπή Γεωργίας για τη διαχείριση ε, του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί και αυτό νομίζω ότι είναι στοιχείο της διαχείρισης της Γεωργίας. Ευχαριστώ. Και πάμε στην τελευταία τώρα ενότητα ερωτήσεων. Αποκλειστική ε, η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη από την ομάδα της που ρωτάει για δεύτερη φορά. Υπάρχει μια οδηγία για τη δυσυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγεία και ιδιαίτερα ε, εναρμόνιση της άσκηση επαγγέλματος. Πρόσφατα ένας γιατρός από ένα κράτος μέλος ε, εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να μιλάει αγγλικά και τελικά ε, έχασε έναν ασθενή του. Πέθανε. και πώς προτίθεστε να ε, κάνετε προτάσεις που θα είναι λογικές, φτηνές και εφαρμόσιμες, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουμε και το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των ασθενών. I have uh, Οφείλω να μελετήσω αυτό το θέμα αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό αφορά περισσότερο το χαρτοφυλάκιο για τη διεθνή αγορά, έτσι, ως προς τη δράση και όχι το δικό μου. Εν πάση περιπτώσει, όταν πρόκειται για τη πτυχή της υγείας και τους επαγγελματίες υγείας και την εγκατάστασή τους, αυτό βεβαίως είναι ε, στο δικό μας ε, τομέα αρμοδιοτήτων και θα πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί για να συνεργαζόμαστε οριζόντια με άλλους επιτρόπους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια των ασθενών. Να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο την αγορά και τα βασικά στοιχεία και τις αρχές ε, της οικονομίας ελεύθερης διακίνησης των επαγγελματιών, αλλά και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικότερο, που είναι οι προδιαγραφές που χρειάζονται για την ασφάλεια των ασθενών. Ah, Ευχαριστώ, κυρία Μισελ Ριβαζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Χαίρομαι γιατί επιτέλους τα φάρμακα επανέρχονται στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και όχι της βιομηχανίας όπως ήταν προηγουμένως. Να επανέλθω στη διαχείριση του εμβολιασμού κατά της γρήπης Α στην Ευρώπη. Υπάρχει επικαιρότητα που δείχνει ότι στις διάφορες χώρες ξοδεύτηκαν άδικα χρήματα για ένα ιό που τελικά δεν ήταν τόσο βαρύς. Αλλά υπάρχουν και θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα διεθνή, τους διεθνείς φορείς και τα, της φαρμακοβιομηχανία. Ρωτώ λοιπόν πώς θα ενισχύσουμε την αντικειμενικότητα και των θεσμικών μας φορέων, είτε αφορούμε αυτό την ΕΦΣΑ, είτε την προστασία από μεταδοτικές ασθένειες σε σχέση με τα φαρμακευτικά εργαστήρια. Αυτό σίγουρα πρέπει να το προσπαθήσουμε, να αξιολογήσουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και να δούμε τι δράση απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ποιοτική υπηρεσία που είναι απαραίτητη για τους ασθενείς. Πρέπει να βρούμε εδώ μια ισορροπία, να εξισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη να έχουμε μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία και την ανάγκη των ασθενών. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε για τίποτα το συμφέρον του ασθενούς, αλλά και μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία είναι προς όφελος του ασθενούς. Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια ισορροπημένη άποψη για ό,τι κάνουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε βεβαίως με την φαρμακοβιομηχανία για την ιεράρχηση της έρευνάς τους. Δεν θέλουμε να τους κατευθύνουμε, αλλά να τους δείξουμε Ποια είναι η άποψή μας, το όραμά μας. για το τι είδους έρευνα περιμένει ο ασθενής. Αλλά αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν πάντως και στους τομείς που αναφέρατε. Κυρία Παρβάνοβα, κύριε Ντάλι, εδώ βρίσκομαι. Δεσμευθήκατε ισχυρά και στις γραπτές σας απαντήσεις να αναπτύξετε πρακτικές κατά της παραποίησης φαρμακευτικών προϊόντων. Έγινε εδώ πολύ ισχυρή συζήτηση για την οδηγία για τα παραποιημένα φάρμακα. Αλλά θεωρούμε ότι αυτή καλύπτει μόνο το 1% των φαρμάκων. Έχετε πρόθεση να αντιμετωπίσετε εις βάθος την, τα παραποιημένα φάρμακα και ιδιαίτερα το εμπόριο μέσω ίντερνετ και το παράλληλο εμπόριο. Απάντηση. Όπως είπα και στις γραπτές μου απαντήσεις στα ερωτήματα σας, θεωρώ ότι η παραποίηση είναι προσβολή του καταναλωτή και κίνδυνος για πολλούς καταναλωτές. Και είναι επίσης μεγάλος κίνδυνος για την προσπάθεια καινοτομίας της Ευρώπης. Δεν είναι κανονικά δύσκολο να ληφθούν βήματα και μέτρα για οτιδήποτε βρίσκεται στον φυσικό κόσμο. Ο φυσικός κόσμος μπορεί να ελεγχθεί και να ε, εποπτευθεί. Και είπα και στις απαντήσεις μου ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσω ότι ό,τι ισχύει για τον πραγματικό κόσμο θα ισχύει και για τον επιγραμμικό κόσμο. Ξέρουμε ότι τα περισσότερα παραποιημένα φάρμακα προέρχονται από ιστοσελίδες. Σήμερα με ελάχιστα χρήματα κάποιος μπορεί να κατασκευάσει μια ιστοσελίδα και να κάνει στην ουσία ό,τι θέλει με αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν είναι όμως εύκολο, είναι πολύ δύσκολο για πολλούς λόγους και για λόγους λογοκρισίας γιατί αρχίζεται να αγγίζεται και θέματα παροχής πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Πάντως θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους επιτρόπους για να αντιμετωπίζουμε την παραποίηση των φαρμάκων. Συμπληρωματικό ερώτημα. Αυτή η πρακτική στην ουσία σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα. Θα συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας που είναι υπεύθυνοι για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και υπάρχουν και άλλα πράγματα που διακυβεύουν την υγεία του κόσμου όπως η ηλεκτρονική ιατρή. Απάντηση. Ναι, όλα αυτά πρέπει να τα προσπαθήσουμε. Είναι σημαντικό να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε και το οργανωμένο έγκλημα και αυτές τις έννοιες των ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως. Αλλά σας είπα, είναι θέμα για το οποίο πρέπει να συνεργαστώ στενά με τους επιτρόπους του κολεγίου. Γιούντιτ Μέρκης. Κύριε Ντάλι, εδώ αριστερά σας. Στα αγγλικά. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού της και αυτό συνδέεται με διάφορες δυσκολίες. Αυτή η δημογραφική αλλαγή όμως δεν αντικατοπτρίζεται ακριβώς ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική δημόσιας υγείας. Εσείς τι θα κάνετε, το θεωρείτε προτεραιότητα, θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρώπη με αυτό το θέμα ή να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών. Και πώς θα θείτε το ίδιο επίπεδο υγείας και περίθαλψης στην Ευρώπη. Και επίσης πώς θα εξασφαλίσετε ο γυράσκον αυτός πληθυσμός να διαφυλάσει παντού την ε, κινητικότητά του. Δεύτερη ερώτηση που απαγορεύεται. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τις μεταφορές ζώων όταν θα πηγαίνουν στα σφαγεία. Ε, the answer is... Η απάντηση είναι ότι βεβαίως και είναι προτεραιότητα η γύρενση. Είναι δημογραφική πραγματικότητα αυτή. Και συμφωνώ ότι όντως δεν αντικατοπτρίζεται ως ε, θα όφιλε στις πολιτικές μας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά στην κατεύθυνση αυτή. Το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού δεν έχει να κάνει μόνο με την περίθαλψη του πληθυσμού που γεννάει. Είναι και τι είδους ζωή χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Να αισθάνονται ότι, πώς να το πω, ότι δεν είναι βάρος στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους. Τα θέματα δηλαδή είναι πολύ ευρύτερα. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα Εντάξει, υπάρχουν ε, ειδικά νοσήματα όπως είναι η γεροντική άνοια, η νόσος Alzheimer κτλ. Όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά πολύ περισσότερο ε, το θέμα είναι ε, ο κόσμος να ζει με τρόπο υγιή για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα είναι εθνική πολιτική ή ευρωπαϊκή πολιτική, Αυτό χρειάζεται μελέτη και θα το μελετήσω, θα εμβαθύνω και τα πάντα θα εξαρτηθούν και από το είδος των λύσεων που χρειάζεται, των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και των βουλειών, είτε είναι αυτές ευρωπαϊκές είτε εθνικές. Και επίσης αυτό συνδέεται και με την κινητικότητα βεβαίως, διότι και πάλι η περίθελψη των ηλικιωμένων είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ασχοληθεί στη Μάλτα ε, το τελευταίο διάστημα, που δύο χρόνια, και δεν είναι μόνο ε, ζήτημα, αλλά είναι και πιεστικό ζήτημα και οπωσδήποτε χρειάζεται ταχεία λύση. Για τις μεταφορές των ζώων μου δώστε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, λίγα δευτερόλεπτα σας παρακαλώ. Για τις μεταφορές των ζώων ε, βεβαίως θα το κοιτάξουμε και αυτό. Ωστόσο, Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι να εφαρμόζεται σωστά η κείμενη νομοθεσία και να γίνει μια επανεκτίμηση ή μια εκτίμηση των ε, όσων εφαρμόζεται. Έχουμε πολύ σαφή γραμμή για το που θέλουμε να πάμε τις μεταφορές στο ζώο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα με το κοινοβούλιο γιατί και η ευημερία των ζώων είναι κάτι που μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει όλους μας. Ευχαριστώ και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θέλουμε να εργαστούμε, αλλά να εργαστούμε γρήγορα ε, γι' αυτό. Και ελπίζω να μας ε, φέρετε σύντομα κάποιους στόχους και για τα δύο θέματα αυτά και για τις μεταφορές των ζώων, αλλά και για κάτι άλλο. Θα σας δώσω το δικό μου χρόνο, αφού δεν προλάβατε να απαντήσετε. Και για κάτι άλλο λοιπόν θέλω να ρωτήσω. Η γύρανση του πληθυσμού θεωρείτε ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και αν ναι, πώς θα το αντιμετωπίσετε και θα το πείτε και στο Συμβούλιο. Ε, We, Ναι, για τις μεταφορές των ζώων θα προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ακούσαμε εδώ όλες αυτές τις ώρες που είμαστε μαζί πόσες προτεραιότητες έχει ο καθένας. Και ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε και κάποια προτεραιότητα στη δράση μας. Με βασική προτεραιότητα ακριβώς την ευημερία των ζώων. Και αυτή. Εγώ δεν είπα ότι είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Είπα ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε και το ζήτημα αυτό. Και αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τις πρωτοβουλίες που θα λάβουμε. Ανάλογα με το ποιο έχει την αρμοδιότητα θα πρέπει να ληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες. Το τελευταίο λόγο θα τον έχει ένας άνδρας ευρωβουλευτής, ο κύριος Ζέμπερ. Καλά, δεν θα είναι ο τελευταίος λόγος κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο υποψήφιος Επίτροπος. Κύριε υποψήφιο Επίτροπε, πώς βλέπετε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και το μοναδικό κοινοβούλιο που αφενός οφείλει κανείς να το λάβει σοβαρά, υπόψη. Από την άλλη μεριά δεν έχει όμως την ε, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, νομοθετικά δηλαδή. Και στην τελευταία θητεία μόνο επτά φορές έκανε χρήση της δυνατότητας αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή να ακούσει μια δική μας πρωτοβουλία όπως είχε τη δυνατότητα να κάνει. Τι θα κάνετε, θα έλθετε εσείς όταν θα είστε πλέον τμήμα ε, μέλος ε, του Συλλογικού Σώματος των Επιτρόπων ε, θα, θα ποιήσετε χρήση αυτής της δυνατότητας που έχετε να δεχτείτε μια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ή ε, μάλλον όχι. Είχα ήδη την ευκαιρία να πω και το ξαναλέω γιατί το πιστεύω ότι η πρόθεσή μου είναι να έλθω να σας δω όσο το δυνατόν νωρίτερα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να ακουστεί η φωνή σας όσο γίνεται νωρίτερα Είπα και πριν ότι προτιμώ να περάσω κάποιο χρονικό διάστημα συζητώντας πολιτική μαζί σας παρά να χάσω χρόνο μετά μαλώνοντας μαζί σας. Θέλω να προχωρήσουμε σε μια μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ε, θέσπιση και άσκηση πολιτικής την οποία ήδη θα έχουμε αρκετά μελετήσει και βασανίσει. Με την έννοια αυτή μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα σας αφιερώσω όλο τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε μαζί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζω ότι και η προκάτοχός μου είχε αναπτύξει τη συνήθεια να έρχεται στο Κοινοβούλιο πριν να προβεί σε οποιαδήποτε σημαντική ανακοίνωση. Και αυτό το βρίσκω θετικό. Όπως είπα και πριν, σας θεωρώ τους εκπροσώπους των ψηφοφόρων σας. Και η αδίποτε ανακοίνωση κάνουμε θα είναι προς τους εντολή σας. Άρα πρέπει να γίνει πρώτα προς εσάς. Ε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ε, εδώ τελειώνει ο χρόνος των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή σας στην ακρόαση από τις ε, Επιτροπές Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Προστασίας Καταναλωτών. Ευχαριστώ και τον κύριο Νταλή για, την, για τις απαντήσεις του. Ε, κάναμε πραγματικά μια ροφή σάρωση του ορίζοντα όλων αυτών των θεμάτων προστασίας ε, καταναλωτών κλπ. Ο κύριος Νταλή έχει 20 ετή πείρα στην πολιτική και αυτό φάνηκε και από τις απαντήσεις του που καμιά φορά ήταν πολύ σύντομες και ακριβείς και συχνά ξανά και ξανά τον επιθύμησε, τον χειροκρότησε η Ντάγμα Ροτ ναι, ναι, Αυτό, πρέπει να, αυτό σίγουρα σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ θετικά αυτά που είπε. Είναι λοιπόν κοινή ακρόαση. Ο Μάλκομ Χάρμπορ της ΙΜΚΟ θέλει και αυτός να απευθύνει λίγα λόγια σε εσά και μετά θα λάβει το λόγο ο ίδιος ο υποψήφιος επίτροπος. Πρώτα, σας ευχαριστώ εξ ονόματος των μελών της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών για τον ε, ευγενικό τρόπο που μας υποδεχθήκατε και η συνεργασία πήγε πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τα 10 μέλη της Επιτροπής μου που έθεσαν ερωτήσεις και ήθελα βέβαια ιδιαίτερα να τονίσω αυτό που ο κύριος Ντάλι απαντώντας στην ερώτηση κ. Κέπχαρτ. Ε, πιστεύω ότι θα είστε όντως ο πρωταθλητής του συντονισμού τη προστασία καταναλωτού μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε καλή συνεργασία και με την κυρία Κούνεβα προηγουμένω και η ο δικό μα ρόλο είναι επίση σημαντικό αφού είμαστε οι θεματοφύλακε του προπολογισμού για την προστασία των καταναλωτών. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μα που ακούσαμε τις ξεκάθαρες αυτές σα και τι διαβεβαιώσει σα για το ότι θα παίξετε τον ρόλο σας ως θεματοφύλακας και χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποίησατε κι εσείς της προστασίας των καταναλωτών. Και σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας αυτές. Γιώργο σας ευχαριστώ και Χάρμπορ. Πέντε λεπτά έχετε κύριε Νταλή για να κάνετε όποια τελικά σχόλια επιθυμείτε. Πρώτα απ' όλα Πρόεδρε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για πολλά θέματα για μένα. Ήδη αρχίζω να κατανοώ το ενδιαφέρον που δείχνει το Κοινοβούλιο για τους διάφορους τομείς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους ιεραρχήσουμε. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε στο μέλλον και τονίζω αυτό το συνεργαστούμε γιατί σας είπα δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει κανένας μόνος του. Η διαχείριση της Ευρώπης είναι βαριά δουλειά και είναι περίπλοκα τα θέματα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Χρειαζόμαστε αυτό το ουράνιο τόξο απόψεων που βρίσκονται σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και αυτό δίνει και προστιθέμενη αξία σε οτιδήποτε κάνουμε στο μέλλον. Ας προχωρήσουμε από κοινού προς το μέλλον λοιπόν και αναμένω τώρα την κρίση σας. Βεβαίως είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για όλα αυτά βεβαίως και θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να εργαστώ σκληρά για να εφαρμόσω πραγματικά την πολιτική πρώτα οι ασθενείς, πρώτα οι καταναλωτές. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταλή. Λήξη στις ακρόσους και στις 4.30 συνεδριάζουν οι συντονιστές στην αίθουσα 1G2.